Right, everybody, welcome. If you could take your seats, please, and then we can um, we can get underway. So I, I apologize uh, for the for the slightly delayed. Καλημέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για την ε, μικρή καθυστέρηση. Είχαμε μία συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών στην άλλη άκρη του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνετε, κάποιες φορές Ε, παρατείνονται αυτές οι συνεδριάσεις. Με τα χαρά σας καλωσορίζω εδώ. Νομίζω πως ε, θα πρέπει τώρα να σταματήσετε τις μεταξύ σας συνομιλίες, παρακαλώ. Εγώ δεν θα κάνω εισαγωγή για να κερδίσουμε χρόνο. Και θα συζητήσουμε το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη που θα είναι η προσφώνηση από τον Χέρμαν Rompuy, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μετά θα ακολουθήσουν ερωταπαντήσεις κάποιες, εισαγωγικές, ε, κάποιες εισαγωγικά λόγια από τον κύριο Γιώζα από την ε, Ουγγρική Εθνοσυνέλευση και ε, αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις έχετε τρία διαφορετικά χρώματα κάρτες. Αν θέλετε να θέσετε ερώτηση στον πρώτη ε, σύνοδο με τον κύριο Φανερομπόη, να χρησιμοποιήσετε το πράσινο χαρτί. Μετά για τη δεύτερη σύνοδο που είναι ο διάλογος μεταξύ βουλευτών να χρησιμοποιήσετε τις ε, θαλασσιές κάρτες και για την απογευματινή σύνοδο την ροζ κάρτα. Για την πρώτη λοιπόν ε, σύνοδο που είναι για σήμερα ε, θα χρησιμοποιήσετε την πράσινη κάρτα αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Με τα χαράς λοιπόν θα δώσω το λόγο στον συνπρόεδρο. Α, αυτό το λέω για τους εθνικούς ευρωβουλευτές. Τα μέλη της ΕΚΟΝ μπορείτε να μου κάνετε και νόημα για, όπως κάνουμε στο Catch the Eye. Ξέρετε πώς θα το κάνετε. Λοιπόν, Ιστβαν. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συμπροεδρεύω ε, στην κοινή συνεδρίαση τη ε, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εισαγωγικά θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, στις 15 Μαρτίου σήμερα εορτάζουμε την Εθνική Γιορτή τη Ουγγαρίας. Το 1848 στις 15 Μαρτίου έγινε η Ουγγρική Επανάσταση ε, και ε, άρχισε να πορεύεται προς την ελευθερία και προς την Ευρώπη ο Ουγγρικός λαός. Και θεωρούμε ότι και το μέλλον μας μας δένει με την Ευρώπη από τότε μέχρι σήμερα. Και προσβλέπουμε πάρα πολύ στην Ευρώπη και από οικονομικής πλευράς αλλά και για τη διατήρηση της δημοκρατίας μας είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και θεμελιώδης να ε, διατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας έχουμε το σύνθημά μας μια ισχυρή Ευρώπη. Και με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που αρχίζει τώρα πιστεύουμε ότι θα κάνουμε βήματα προς τα εμπρός για την ενίσχυση της συνεργασίας. Επίσης θα ε, θέλαμε σε γενικές γραμμές να θέσουμε τις βάσεις για την ευρωπαϊκή οικονομική ε, δραστηριότητα, πρώτα τα γενικά δηλαδή τις αρχές και μετά να περάσουμε στις λεπτομέρειες. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη είναι πιο ισχυρή όντας ενωμένη και ολοκληρωμένη και ενοποιημένη και αυτό ε, δίνει πλεονεκτήματα για την αγορά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν. Επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα συνεισφέρει πάρα πολύ στη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ε, ο κύριος Φανρόμπαε, αλλιώς να συνεχίσω εγώ να μιλάω μέχρι να έρθει. Σας έλεγα λοιπόν ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο μας ε, προσφέρει νέες ευκαιρίες τώρα. Ευκαιρίες έτσι ώστε μετά από διαβουλεύσεις να μπορούμε να διαμορφώνουμε αυτό το πρόγραμμα οικονομικής δράσης στην Ευρώπη, το οποίο πηγαίνει πολύ περισσότερο από τη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα. Μπορεί ορισμένα κράτη-μέλη να θεωρούν ότι περιορίζεται έτσι ε, το περιθώριο χειρισμών που είχαν μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ περισσότερες οι ευκαιρίες από τους περιορισμούς. Η Ευρώπη για να πετύχει στη διαχείριση της κρίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει αποφασιστικά βήματα προς την εκτέλεση των στόχων της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την καινοτομία. Χρειάζεται μια Ευρώπη πραγματικά ολοκληρωμένη. Αρχίζει μια δεκαετία πάρα πολύ σημαντική πλέον. Δεν θα πρέπει να καθυστερούμε απέναντι στην οικονομική κρίση. Δεν δικαιολογούνται πλέον ολιγορίες και παλινοδίε. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε και διαρθρωτική κρίση στην όλη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού ε, συστήματος και στις χρηματαγορές. Και αν μπορέσει η Ευρώπη να είναι στην αιχμή του δόρατος, της αλλαγής των συστημάτων, της αύξησης διαφάνειας, αυτό δεν θα είναι μόνο προς όφελος της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Και θα βελτιωθεί και η διαφάνεια του παγκοσμίου χρηματοοικονομικού συστήματος. Τελειώνω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, Σάρων, που μου δώσετε το λόγο. Θα δώσω μέσα το λόγο στον κύριο Φαν Ρομποϊ, που μόλις κατέφτασε. Ευχαριστώ. Thank, thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά καλωσορίζω τον Πρόεδρο Φαν Ρομποϊ που θα μας προσφωνήσει. Πράγμα το οποίο θα ακολουθηθεί από ερωταπαντήσεις. Χαιρόμαστε πολύ που είχατε το χρόνο να έρθετε να μας ε, κάνετε αυτή την προσφώνηση, ενώ είστε τόσο απεσχολημένος. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, και εθνικοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα βλέπω συχνά. Έχουμε πάρα πολύ ζωντανές συζητήσεις στην Ολομέλεια. Εγώ ως πρώην Εθνικός Βουλευτής και ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής αισθάνομαι πάντα χαρά και ευχαρίστηση να έρχομαι στα παλιά μου λιμέρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον καιρό λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις για να βελτιώσει την κοινή μας οικονομική διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς και της Ευρωζώνης. Για το λόγο αυτό θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός Ε, ότι τα κοινοβούλια που ενέχονται άμεσα έχουν κάνει κτήμα τους αυτή την προσπάθεια και την έχουν ενστερνιστεί. Θα πρέπει να αξιοποιείτε κάθε ευκαιρία ε, που έχετε να εκφράζετε την απόψή σας και να λαμβάνονται οι απόψεις σας πραγματικά υπόψη. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή ευκαιρία και συζήτηση. Εισαγωγικά θα ήθελα να μιλήσω ε, λίγο για το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Περίεργο είναι αυτό το, ως όρος και να σας ενημερώσω επ' για τις πιο ε, πρόσφατες εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταθερά βγαίνει από την οικονομική κρίση. Ας δούμε μερικά θεμελιώδη στοιχεία. Τα οικονομικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης στο σύνολό της παραμένουν υγιή, χαμηλή, ε, χαμηλός πληθωρισμός, ε, πληρωμών τρέχουσών συναλλαγών ισορροπημένο σε σχέση με άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές των παγκοσμίων πραγμάτων. Και σύντομα θα επανέλθουμε σε οικονομική ανάπτυξη μετά την χρηματοοικονομική κρίση. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουμε πρόβλημα στα θέματα δημοσίου χρέους. Η κρίση έδειξε πώς τα προβλήματά μας μπορούν να εξαπλωθούν από μία χώρα και να επηρεάσουν και όλες τις υπόλοιπες με ταχύτητα και μέγεθος που πολλοί δεν θεωρούσαν ε, δυνατό. Πέρυσι κατέστη σαφές ότι χρειαζόμαστε επιγόντως να μάθουμε ε, ακριβώς, να εξάγουμε διδάγματα από αυτή την εμπειρία. Οι πρώτες λοιπόν Συνεπής και τα πρώτα συμπεράσματα εξήχθησαν στη λεγόμενη Task Force, ομάδα εργασία για την οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα επεξεργαζόμαστε ένα δεύτερο σύνολο συμπερασμάτων και συζητούμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωζώνη την περασμένη Παρασκευή και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε επίπεδο πλέον 27 στα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και να κάνουμε μια στροφή. Ε, είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία μας απασχολούν. Το κάθε ένα ξεχωριστά μπορεί να είναι μικρό, αλλά συνολικά όλα σημαίνουν μεγάλη αλλαγή, ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εμεί οι Ευρωπαίοι διαχειριζόμαστε την ολοκληρωμένη, την ενοποιημένη μας οικονομία, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Το βασικό μου μήνυμα είναι το εξής. Όλες οι αποφάσεις μας θα χρειάζονται να βρίσκουμε μια νέα ισορροπία για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μια ισορροπία μεταξύ της κοινή ευθύνη, που μπορείτε να την ονομάσετε και αλληλεγγύη αν θέλετε, και της μεμονωμένη ευθύνη κάθε κράτου ξεχωριστά. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο σήμερα συζητάτε εδώ, είναι ε, τμήμα αυτή τη εξίσωση. Από την πλευρά τη αλληλεγγύη ελήφθησαν ε, επίκαιρες δράσεις, ο προσωρινός μηχανισμός σταθεροποίησης, τα πακέτα για την Ελλάδα και την Ιρλανδία και ε, σχέδια για να γίνει ο μηχανισμός αυτός μόνιμος. Σε ό,τι αφορά τη μεμονωμένη ευθύνη, αυτό σημαίνει σκληρά μέτρα και επίγοντα ε, εσωτερικά μέτρα σε πολλές χώρες. Τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα, όχι μόνο πολιτικά βέβαια. Ας πούμε, ο μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας 500 δισεκατομμύρια ενδεχομένω δανείων που εγγυώνται τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτά είναι τεράστια ποσά, οπότε είναι φυσικό οι διαπραγματεύσεις να ε, συνδέονται με επιπλέον υποσχέσεις και δεσμεύσεις για να περιοριστούν τα ποσά αυτά. Και μεταξύ αυτών είναι δύσκολα μέτρα λιτότητας και μεταρρυθμίσεων σε χώρες με μείζωνα ελλείμματα. Οι πολιτικοί περιορισμοί ε, κατέρωθεν και τα προβλήματα είναι αρκετά σοβαρά, όπως τα γνωρίζετε. Τα κράτη χρειάζεται να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και χρειάστηκε να λάβουν θαραλέες αποφάσεις. Επιτυχάνουν στην προσπάθεια αυτή. Το ίδιο ίσχυσε και για κυβερνήσεις οι οποίες χρειάστηκε να πείσουν τα κοινοβούλια τους και την κοινή τους γνώμη να μπουν σε δανειακές συμβάσεις, βεβαίως με πάρα πολύ αυστηρούς όρους. Για εκείνους ε, είναι επίσης υψηλό το διακύβευμα. Και στις δύο περιπτώσεις η Ευρώπη ούτε ήταν ούτε είναι δημοφιλής. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας ε, εμποδίσει από το να δράσουμε και υπέρ της αλληλεγγύης και υπέρ της ευθύνης. Ας μην λησμονούμε ότι αν δεν λαμβάναμε αυτές τις αποφάσεις η κρίση θα ήταν πολύ χειρότερη και είναι προς όλων να διατηρηθεί η σταθερότητα της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Επίσης, αυτό ε, δίνει και μεγάλη ευθύνη στα εθνικά κοινοβούλια. Ο μηχανισμός σταθερότητας θα χρειαστεί ομοφωνία, ας πούμε, όλων των κοινοβουλίων. Και η δική σας συμμετοχή δίνει την απαραίτητη νομιμότητα στην προσπάθεια αυτή. Και επίσης η φωνή σας θα επηρεάσει όλους τους υπολείπους, γιατί εσείς δεν αποφασίζετε μόνο για τη δική σας πατρίδα, αλλά για όλες τις χώρες μας. Στο μέλλον, για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θέλουμε να περιορίσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο να ξανασυμβούν τέτοια προβλήματα. Και επιτρέψτε μου σας αναφέρω τρία βήματα ε, και σκέψεις αλλά και δράσεις Πάντα με μεγαλύτερη ατομική ευθύνη. Πρώτον, ανακαλύψαμε και μάλιστα με το σκληρό τρόπο ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που στην αρχή είχε σχεδιαστεί με κάποιο τρόπο δεν ήταν αρκετά ισχυρό. Το σύμφωνο αυτό έχασε πολύ από την ισχύ του όταν το 2003 παραβίασαν τους κανόνες δύο μεγάλες χώρες. Όταν ομολόγησε η Ελλάδα έλλειμμα που έφτανε κοντά στο 15% του ΑΕΠ στα τέλη του 2009, τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Η ομάδα ε, ε, δράσης για την οικονομική διακυβέρνηση, της οποίας προείδρευσα πέρυσι, ε, πρότεινε να ισχυριοποιηθεί, να αυστηροποιηθεί το σύμφωνο με νωρίτερες κυρώσεις, πιο αυστηρές και πιο προσιλωμένες στο δημόσιο χρέος. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν να λάβουν κάποια μέρα, το, μέτρα το Μάρτιο, βεβαίως σε συναπόφαση μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι το, Ιούνιο, μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκτός λοιπόν από την ενίσχυση αυτού του συμφώνου σταθερότητα, έρχεται να προσθεθεί και το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό δεν είναι όπως ισχυρίζονται ορισμένοι μία άσκηση ε, όπου οι Βρυξέλλες ε, επισέρχονται στα, εσωτερικά των κρατών, παρεμβαίνουν και τους λένε πώς να καταρτήσουν τον προϋπολογισμό τους. Όχι, αυτό παραμένει ε, στα χέρια των κρατών μελών και είναι βασικό στοιχείο κάθε κράτους και κάθε δημοκρατίας. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με κάποιους στόχους, δημοσιοοικονομικούς, μακροοικονομικούς και θεματικούς. Σκεφτείτε τη στρατηγική για το 2020. Οι εξελίξεις λοιπόν εδώ ε, κατευθύνονται στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια πορεία. Και αυτό είναι εκ των όνων για τις χώρες του ευρώ. Η οικονομική δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης είναι προς όφελος όλων. Τα κράτη-μέλη θα καταρτίζουν τα προγράμματά τους, εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και για τη σταθερότητα ή τα προγράμματα σύγκλησης του προπολογισμού. Θα καταρτίζουν από τα κράτη τα προγράμματα αυτά, τα οποία θα ε, αξιολογεί η τα προγραμματα συγκλησης του προπολογισμου θα καταρτιζουν λοιπον τα κρατη Επιτροπή και στη συνέχεια η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο, στα κράτη-μέλη δηλαδή, ειδικέ συστάσεις και γνώμες ανά χώρα για τα εκάστοτε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και ε, τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκληση. Οι συστάσεις αυτές που εγκρίνονται από το Συμβούλιο θα λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των σχεδίων προπολογισμών για το 2012. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και για σας, διότι μπορεί να φέρει μια ευρωπαϊκή διάσταση και στις εθνικές συζητήσεις σας. Γιατί σήμερα λείπει πάρα πολύ συχνά αυτό το στοιχείο. Για παράδειγμα, αν μια κυβέρνηση επιλέξει να μην ακολουθήσει κάποια σύσταση, φέρει μπορεί η Βουλή να το ζητήσει στη χώρα. Και αν δεν το κάνουν αυτά τα κυβερνώντα κόμματα, μπορεί να το κάνει η αντιπολίτευση. Και εσεί ως Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχετε ρόλο κλειδί πρωταγωνιστικό να διαδραματίσετε εδώ. Βεβαίω, το περιεχόμενο του προπολογισμού, τι επιλέγει μια χώρα να δαπανάει, να φορολογεί, παραμένει εθνική υπόθεση και απόφαση. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο βήμα κυρίες και κύριοι όσον αφορά τη βελτίωση της αίσθηση της ατομικής ευθύνης. Αυτό προέκυψε με την ε, διαπίστωση ότι ορισμένοι προπολογισμοί δεν αρκούν για την εγγύηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι άλλο ένα μήνυμα της κρίσης. Στην πρώτη δεκαετία του ευρώ, με μεγάλα επιψηλά επιτόκια και σταθερότητα στην Ευρωζώνη, η απώλεια ανταγωνιστικότητα κατέστη αόρατη. Όμως οι φούσκες, οι, η υπερμεγέθεις των τραπεζών παραβλέφθηκαν και γι' αυτό τώρα ε, δημιουργούμε ένα είδος μακροοικονομικής εποπτείας ε, που θα παρακολουθεί τέτοιου είδους κινδύνους και ανισορροπίες. Αν το είχαμε αυτό ήδη στο ενεργαλειοθήκη μας εξ αρχής ε, του ευρώ, πολλά πολλά προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί. Και αυτό μας οδηγεί στο πιο πρόσφατο βήμα που αφορά την αυξανόμενη δέσμευση των χωρών της Ευρωζώνης να σύρουν τα διδάγματα του κοινού νομίσματος. Ξέρουμε πως υπάρχει ένα σύστημα όπου έχουμε οικονομική ένωση χωρίς επαρκή οικονομική ενότητα. Ως αποτέλεσμα της κρίσης λοιπόν οι κυβερνήσεις λένε πια ότι πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Για μένα αυτό είναι εξέλιξη κλειδί προφανώς ε, δεν θα υπάρξει μια ξαφνική μετάβαση σε ευρωφορολογία, ευρωομόλογα κτλ. Μπορεί να λυπούμεθα γι' αυτό, αλλά πολιτικά αποκλείεται για την ώρα από όλα τα κρατημέλη. Θα πρέπει αυτό λοιπόν να το δεχτούμε. Φορολογική πολιτική και σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αγορά εργασίας παραμένουν ευθύνες ε, των εθνικών δημοκρατιών της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα το ευρώ είναι και παραμένει το κοινό μας νόμισμα. Αντί λοιπόν να κεντροποιούμε τις πολιτικές και τα μέσα και αντί να μην κάνουμε τίποτα, μιλάμε για συνδυασμένες ενέργειες, για συντονισμό των εθνικών πολιτικών. Και πάλι πρόκειται για ανάληψη των ευθυνών από τις μεμονωμένες χώρες μέλη για το σύνολο της Ευρωζώνης. Αυτή η πεποίθηση πως οι χώρες Ευρωζώνης πρέπει να κάνουν περισσότερα είναι τώρα μια πεποίθηση που μοιράζονται όλοι οι ηγέτες της Ευρωζώνης. Στην περασμένη σύνοδο της Ευρωζώνης, την περασμένη εβδομάδα, συμφωνήσαμε για ένα σύμφωνο, όπως το αποκαλέσαμε, για το ευρώ. Εντοπίσαμε πέντε κύριους στόχους. Ανταγωνιστικότητα, ανταγωνιστικότητα των μισθών, απασχόληση, βιώσιμη δημόσια οικονομία και τραπεζικά συστήματα, συντονισμός φορολογικός και οικονομική σταθερότητα. Με βάση κάποιου δείκτε θα εντοπίσουμε τι χώρε που πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένε ενέργειε. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία και θα εκτιμά την εφαρμογή των μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν για να συμμορφωθούν προ τα... τι προδιαγραφέ. Το ίδιο ίδια προσέγγιση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τώρα, πώ θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίε θα είναι εθνικό θέμα. Αλλά η ανάλυση και ο εντοπισμό των προβλημάτων που επηρεάζουν όλου θα γίνει από κοινού. Επιπλέον, δεν θέλουμε μόνο να κεντροποιήσουμε τις διαδικασίες στις Βρυξέλλες, πρόκειται για πολιτική δέσμευση. Οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων θα ανακοινώσουν μέτρα υπό το σύμφωνο για το ευρώ, το οποίο, το οποίο θα τα εφαρμόσουν εθνικά. Αν φυσικά συμφωνήσουν τα κοινοβουλιά τους. Άρα λοιπόν, εκτός από την πίεση της αγοράς και εκτός από τις, ε, την υφιστάμενη θεσμική πίεση, δηλαδή σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξης μακροοικονομικής ε, υποπτίας, τώρα θα έχουμε ισχυρότερη πίεση από τους ε, υπολείπους της Ευρωζώνης. Έτσι, οι συμμετέχοντες στο Ευρωσύμφωνο θα θα δεσμευθούν και πολιτικά. Ορισμένοι λένε πως αυτό δεν είναι αρκετά δεσμευτικό, ενώ άλλοι θεωρούν ότι ένα τέτοιο σύμφωνο θέτει σε κίνδυνο το κοινωνικό μας πρότυπο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι τα περισσότερα μέτρα χρειάζονται στο εθνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, τα συνταξιδοτικά συστήματα και το πώς αυτά θα είναι βιώσιμα και πώς η οικονομία θα είναι ανταγωνιστική. Οι τεχνικές των οικονομικών, της οικονομικής διακυβέρνησης πιέζουν τα κράτη-μέλη, διότι έχουμε κοινά συμφέροντα. Το ευρώ. Αυτό δεν κάνει την Ευρώπη πολύ δημοφιλή, το έχω ήδη πει. Αντιθέτως η Ευρώπη είναι μια, μια αντιπαθητική ιδέα. Φυσικά είναι κατανοητό όσοι ε, μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα να κάνουν περισσότερα από κοινού. Από την άλλη πλευρά, ε, οικονομικά και πολιτικά θα είμαστε όλοι πολύ συνδεδεμένοι. Οι ευκαιρίες ε, επίσης επηρεάζουν τα κράτη. Σκεφτείτε το σύνδεσμο ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Επιπλέον πολύ ακόμα θα μπουν στο ευρώ στα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, οι συνάδελφοι που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη θα ανακοινώσουν αν θέλουν να συμμετέχουν στο Ευρωσύμφωνο ή όχι. Για να κλείσω, κύριε και κύριοι, το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης φαίνεται ένα πιο ανθυρό η συλλογική και η ατομική ευθύνη καθενός για το ευρώ είναι πιο εξασφαλισμένη και η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη είναι καλύτερη από ό,τι αναμενόταν. 1,6 ε, φέτος και 2,0 για τον επόμενο χρόνο προβλέπεται. Να προσθέσω όμως πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν απαραμέλησε το θέμα της δομής της οικονομικής ανάπτυξης και γι' αυτό θεσπίσαμε αυτή τη στρατηγική 2020 Αναπτύξαμε και μια στρατηγική για την ενέργεια και την καινοτομία και γι' αυτό και η Κομισιόν ξεκίνησε το «In πράξη» της ενιαίας αγοράς. Έπειτα, η πολιτική αποφασιστικότητα είναι σταθερή στο η και στο μυαλό των ε, ηγετών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το μέλλον είναι ευρωπαϊκό. Είναι ένα πολιτικό γεγονός το οποίο πρέπει πάντοτε να το έχουμε υπόψη μας. Ορισμένοι ξέρω πως πιστεύουν πως δεν θα τα καταφέρουμε, ωστόσο διαρκώς έχουμε ε, λάβει δύσκολες αποφάσεις τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η αγάπη, όπως λένε οι Γάλλοι, αποδεικνύεται έμπρακτα. Και όπως λένε και οι Άγγλοι, το αν είναι καλό ένα γλυκό το βλέπει κανείς τρώγοντάς το. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στις αποκρίσεις. Έξι πράσινες κάρτες έχω δει από εθνικούς βουλευτές και τέσσερις ευρωβουλευτές που ζήτησαν το λόγο από την Επιτροπή μας που ε, μου έκανα νόημα. Λοιπόν, αν μιλήσετε πάνω από τρία λεπτά δεν θα προλάβουμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, να σας πω τα ονόματα. Από το Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, χώρες θα σας πω, για να μην λέω λάθος τα ονόματά σας, είναι πιο εύκολο. Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Ρουμανία από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου Περβάν Περές και ο Συγκαρσία Μαργάιου, Σοφή και ο Μιγγέλ Πόρτας. Λοιπόν, επειδή κινδυνεύουμε να έχουμε επικαλύψεις στις ερωτήσεις, προτείνω να τις ομαδοποιήσουμε και μετά θα ζητήσω από τον πρόεδρο Βανόμπο να απαντήσει συλλογικά. Λοιπόν, Κρίστοφ Μάτσνερ από την Αυστρία, παρακαλώ. Δεν ξέρω που κάθεστε, δεν σας βλέπω. Yes, the floor is yours. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φανρόμποε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σαφή περιγραφή των δυσκολιών για το επόμενο διάστημα για όλα τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ε, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες ε, θεσμικές προϋποθέσεις. Οι χώρες ε, που δεν το έχουν αυτό ε, το χρειάζονται. Δηλαδή συντονισμένη προσπάθεια, συντονισμένη δράση. Γιατί κάθε 15 μέρες ε, ξυπνάμε με την αγωνία τι θα γίνει με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σπρέτς στις χρηματαγορές. Με τελευταίο παράδειγμα την Πορτογαλία που εκτοξεύτηκαν τα επιτόκια. Και το ερώτημα είναι, παραμένει αηφόρο αυτό, δηλαδή ο συντονισμός και μόνο οι μηχανισμοί διάσωσης ε, με τόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά αρκούν από μόνα τους. Γιατί έχουμε ζήσει και την κρίση στην Ασία το 1998 και ο καθένας διερωτάται γιατί εσείς οι Ευρωπαίοι είστε τόσο συγκρατημένοι και τόσο επιφυλακτικοί ιδιαίτερα απέναντι στις χρηματαγορές. Και νομίζω ένα βουλευτής δικαιούται να κάνει αυτή την ερώτηση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση ε, ικανοποιητική. Εξακολουθεί η κερδοσκοπία να επιτίθεται ανοιχτά σε μεμονωμένα κράτη-μέλη πέρα από τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και παραγνωρίζοντάς τις. Πώς είναι δυνατόν με CDS να κινούνται τόσα πολλά από εσά τα παράγωγα και ε, δεν ε, επιτρέπουν ε, όχι μόνο να δανείζεται κανείς σε λογικές τιμές αλλά προχωρούν και σε προφητείες για θέτηση πληρωμών. Αυτά τα credit default swaps. Ε, τι στοιχήματα είναι αυτά. Δηλαδή ε, μπορεί κανείς να ποντάρει σε ένα ε, άλογο που ξέρει ότι δεν τρέχει, ότι είναι άρρωστο και πληγωμένο και δεν πρόκειται να τερματίσει ποτέ. Θα πρέπει να απαγορεύονται αυτά τα, τα στοιχήματα. Αρχίζουμε να συζητάμε για εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, μετά θα πάμε στο 1 δισεκατομμύριο και μετά δεν θα έχουμε χρήματα. Και θα αρχίσουν σιγά σιγά να πυροβολούν ε, με μονομένες χώρες. Σε 217% ε, που έχει εξωτερικό χρέος η Ιαπωνία δεν τόλμησε κανείς να της επιτεθεί κερδοσκόπος. Και το βλέπουμε σήμερα ακόμα μετά από 13 χρόνια δεν τολμάει κανένα μεγάλο hedge funds να επιτεθεί στην Ιαπωνία με CDS. Τα λέω αυτά πρόεδρε ε, για να μου πείτε αν έχουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, αν θα τις δούμε, όχι μόνο παθητικές, ενεργητικές, ε, να ε, υποστηρίξουμε και να υπερασπιστούμε το κοινό μας νόμιζα με το ευρώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παπανδρέου από την Ελλάδα. Papandreou. Η κυρία Παπανδρέου παρακαλώ όταν είπατε κάτι. Okay. Thank ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρομπάη για την παρουσίασή του και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να έχουμε αυτές τις δυνατότητες ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ε, δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Ρομπάη. Είπε ότι η Ευρώπη ανακάμπτει και βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ ε, θετικό και ότι χρειάζεται μια νέα ισορροπία μεταξύ οικονομικής και νομισματικής ένωσης και από εκεί και πέρα ανέφερε διάφορα μέτρα και βήματα τα οποία έχουν ε, πάρθει για να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα ισορροπία. Θεωρείτε, κύριε Ρομπάη, ότι ο συντονισμός, ο οποίος είναι απαραίτητος, δεν τον αμφισβητεί κανείς, και οι ποινές, που και αυτές είναι απαραίτητες, αλλά από μόνες τους αρκούν για την δημιουργία του, ε, της Ευρωμένης Ευρώπης δεν ίσως θα έπρεπε να έχουμε και κάποιους μηχανισμούς αποτρεπτικούς ε, καινούριων κρίσεων, γιατί για να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και τους Ευρωπαίους πολίτες. Και όπως είπατε και εσείς, η Ευρώπη δεν είναι και τόσο συμπαθής σήμερα. Ε, και πώς θα ήταν συμπαθής όταν σε αυτή την οικονομική κρίση, η οποία κατά γενική ομολογία. Προήλθε από τις χρηματαγορές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν ότι αυτοί φέρνουν την κύρια ευθύνη και την κύρια, ε, και την κύρια ποινή. Παίρνετε, τα μέτρα είναι για περιορισμό μέτρα λιτότητας για όλες τις χώρες και βεβαίως πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μπορεί όμως ένα μοντέλο ανταγωνιστικότητας να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική κατάσταση της ε, κάθε χώρας. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της ανεργίας που αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως είναι ευθύνη μας να μην κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές τεράστια χρέη και ελλείμματα. Είναι όμως επίσης ευθύνη μας να μην κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές τεράστια ελλείμματα σε θέματα παιδείας, υγείας και υποδομών. Και φοβάμαι ότι με την πολιτική που ακολουθούμε ε, οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν μόνο το βάρος των ελλημάτων των δημοσιονομικών, αλλά θα έχουν και μία Ευρώπη με λιγότερες δυνατότητες. Ίσως πάμε σε μια χαμένη ε, νέα ε, γενιά. Μετά από δύο χρόνια. Ε, τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I've... Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο-ένα είναι οι, εθνικοί βουλευτές με την εικόνα. Η Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε ότι εδώ είμαι. Ε, εγώ με την ιδιότητα της εισηγήτριας εδώ στο Κοινοβούλιο για το εξάμεινο του Ευρωπαϊκού καταλαβαίνετε ότι το σημαντικότερο θέμα είναι η θέληση να δημιουργήσουμε μια στρατηγική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το G20. Αν δεν θέλει κανείς αυτό το εξάμεινο να ε, να μην, να έχει, μην πετύχει, θα πήγαινε κατανοητό ότι ε, ήδη είχαμε κάνει μια προσπάθεια να ενταχθεί αυτό το εξάμεινο στην οικονομική ανάπτυξη ε, και οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι περισσότερο ακαδημαϊκή και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν κοιτάω το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση, δέχεστε μια αξιολόγηση όσον αφορά τις δαπάνες της δημόσιες, ζητάτε ε, βλέπετε το θέμα των συντάξεων με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Διότι μέχρι τώρα είχαμε απόδειξη ότι απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνα. Όταν έχουμε με ασφάλειες, τράπεζες, με τις μηχανισμούς που ξέρετε πολύ καλά που ισχύουν, ξέρετε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά την αξιολόγηση. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν αν θέλουμε δηλαδή να δούμε την επιτυχία στο βάθος, να καταλάβουμε πώς γίνεται, πώς είναι, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε τις δημόσιες δαπάνες στο μέλλον. Και επίσης, όταν βλέπω τον τρόπο της Επιτροπής όσον αφορά το σύμφωνο για το ευρώ, έχουμε ένα οδοστρωτήρα που διαπιστώνουμε, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλα τα κοινωνικά μοντέλα όποιο και να είναι το σημείο κίνηση για οποιοδήποτε κοινωνικό μοντέλο. Μήπω στην αξιολόγηση ε, που θα γίνει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε να κάνουμε μια διαφοροποιημένη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλέ πτυχέ, Διότι υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως θα πρέπει δηλαδή να σεβαστούμε αυτά τα διαφορετικά μοντέλα και να δούμε πώ μπορούν αυτά να εμπλουτίσουν την πολιτική μα. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ και ερχόμαστε τώρα στον κύριο Καραβάλιο από την Ιταλία. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου, αυτή την ε, περίοδο η Γερουσία συζητά την ε, νομοθεσία σχετική με την δημόσια οικονομία που είναι ε, απαραίτητη νομοθεσία για να τροποποιήσουμε τις πολιτικές μας για το επόμενο εξάμεινο και αυτό θα εγκριθεί πριν από την έναρξη της 30 Απριλίου. Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν πιο αυστηρούς νόμους για την κάλυψη και κυρίως την πρόβλεψη στην φάση οικονομικού προβλήματος προγραμματισμού από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Αυτό θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να εκφράσει κατευθύνσεις για τους στόχους που και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις, πριν τις 30 Απριλίου. Επίσης συζητήσαμε για τη σκοπιμότητα πιο ευθυρών ε, νομοθεσιών σε σχέση με τον περιορισμό του ελλείμματος. Ωστόσο, αποφασίσαμε να περιμένουμε ε, την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την διακυβέρνηση πριν να εισάγουμε νέες δεσμεύσεις. Η βασική δυσκολία που προέκυψε στη διαδικασία προσαρμογής εφαρμογή της διαδικασίας της για το νέο εξάμεινο ήταν ότι είχαμε πολύ περιορισμένο χρόνο για τον ε, οικονομικό προγραμματισμό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε αξιόπιστους στόχου, θα πρέπει να έχουμε ε, αξιόπιστα στοιχεία τα οποία αφορούν το, το καθάριστο εγχώριο προϊόν για το προηγούμενο χρόνο και είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο. Έχουμε λιγότερο από 30 μέρε δηλαδή για να καθορίσουμε την εθνική μα οικονομία. την πολιτική μας για την εθνική οικονομία οικονομία για τον επόμενο εξάμεινο. Είναι σημαντικό και για τους μακροοικονομικούς στόχους, γιατί είδαμε ότι το παλιό σύμφωνο σταθερότητας που βασιζόταν μόνο σε δεσμεύσεις του εθνικού προπολογισμού δεν λειτουργήσε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχουμε από το Βέλγιο τον κύριο Βαντεμπρούκ. Εδώ μπροστά. Yeah, thank you well. Uh- ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στο Βελγικό Κοινοβούλιο έγινε εκτενέστατη συζήτηση μετά από μια ερώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ήταν ευρύτατη συνένεση τελικά. Όλα τα δημοκρατικά κόμματα συμφώνησαν ε, για ε, να δώσουμε τις ίδιες απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Θέλω να τονίσω ότι οι συμφωνίες που γίνονται για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Και Επίσης επιθυμούμε να είναι πάρα πολύ αυστηρή η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Το τονίσαμε αυτό. Επίσης στο Βελικό Κοινοβούλιο υπάρχει συνένεση για τις προτάσεις που από ό,τι ακούω είναι αντιφατικές επίμαχες. Δηλαδή ευρωομόλογα που να χρηματοδοτούν όμως διευρωπαϊκά έργα διασυνοριακά, σε αυτό συμφωνούμε εμείς. Και υπάρχει πραγματικά ευρεία συνένεση από αυτού για τα ομόλογα για τα έργα. Θα ήθελα όμως επ' να σας πω ότι υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα ε, και θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο Φαρόμπαε. Συμφωνώ απολύτως κανονικά με την άποψη που λέει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την αντιπαραγωγική πόλωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποδιοποιημένη πομπαίο τράγο για μέτρα που έτσι κι αλλιώ θα πρέπει να πάρουμε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των ε, κρατών μα το κράτο πρόνοια. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Φαρόπα. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε μία αντιπαραγωγική πόλωση. Για να γίνει αυτό όμω, για να μην στραφεί ο κόσμο κατά τη Ευρώπη, θα πρέπει να είμαστε διαβεβαιωμένοι και σίγουροι ότι η υποκείμενη στρατηγική στην οποία εδράζεται το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ισορροπημένη και αρκετά ευρεία. Γιατί το λέω αυτό. Είναι μεγάλη στόχη για τη στρατηγική του 2020. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αποφύγουμε όμως, δηλαδή από πλευράς μεθόδων και ε, προσέγγισης, πώς μπορούμε λέω, να αποφύγουμε τους επόμενους μήνες οι απογοητεύσεις που έχουν δημιουργηθεί από τη ε, στρατηγική της Λισαβόνας να ε, επαναληφθούν. Ας πούμε, παιδεία, έρευνα, ανάπτυξη, εργασία, κοινωνική συμπερίληψη. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν πλήρης αποτυχία και θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε εντελώς. Δεν είμαι μεταξύ των υπερσκεπτικιστών. Ε, Έχω πιο ισορροπημένη άποψη. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε μία αξιολόγηση για τα θέματα τα κοινωνικά και της ε, εργασίας και της απασχόλησης. Λοιπόν, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μία σωστή και πλήρη συμμόρφωση και εφαρμογή αυτών και αν τα κράτη δεν επιτυχάνουν ας πούμε τους στόχους ε, για τα πανεπιστήμια, για την έρευνα και ανάπτυξη ή για την κοινωνική συμπερίληψη θα πρέπει να δέχονται και αυτά συστάσεις. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Uh, Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα. Ο Χωσέ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέει Κύριος Σκαρίγα, Πογέ. Καλώς ορίσατε κύριε Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο εδώ έχει ορισμένες εμονές και μία από τις εμονές αυτές είναι να μπαίνει σε ένα συστηματικό σύνολο αυτό που συζητούμε τώρα, τα έξι μέτρα δηλαδή για τη διακυβέρνηση και οι προτάσεις που συζητώνται εκτός Κοινοβουλίου, όπως έγινε στη Σύνοδο Κορυφής στις 11 Μαρτίου. Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι υπάρχει δεν υπάρχει επικάλυψη ε, με την πρόταση για ε, το σύμφωνο για το ευρώ, για την ανταγωνιστικότητα και τις δημοσιονομικές ε, πολιτικές. Δεύτερον, στο μηχανισμό διάσωση αποφασίστηκε από το 2013 σημειοτοχή και του ιδιωτικού τομέα. Πώς θα αποφύγουμε το καθεστώς που επιβάλλεται στους τίτλους που θα εκδοθούν από το 2013, πώς θα αποφευθεί αυτό να επηρεάσει, να μολύνει τίτλους που έχουν εκδοθεί πριν το 2013. Επίσης, το πακέτο της διακυβέρνησης πώς εντάσσεται και πώς συνάδει με το μηχανισμό διάσωσης. Γιατί εγώ τι προτείνω. Η πολιτική απάντηση ε, των κρατών ε, στις συστάσεις που θα τους γίνονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, όταν κρίνουμε ε, ε, το χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Και για τις τράπεζες και τη ρύθμισή τους. Τι γίνεται με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ποιοτική διαφορά του δημόσιου χρέους. Ε, ανεξάρτητα από το χρέος σήμερα, ανεξάρτητα από τη φύση του και το spread, το χρέος δεν καταναλώνει δημόσιο χρήμα. μπορεί να υποβαθμιστεί το χρέος των κρατών που κινδυνεύουν και δεν ε, συμμορφώνονται με τις συστάσεις. Και αν αποφάσισε το Συμβούλιο ότι μπορεί να αγοράσει στην πρωτογενή αγορά δημόσιο χρέος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα εμπόδιο να μιλήσουμε για κοινά ομόλογα, για τα ευρωομόλογα στη συζήτηση που θα έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, πάντα με την ευθύνη του καθενός. Εσείς συμφωνείτε, Πρόεδρε, ή διαφωνείτε με όλα αυτά Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ερχόμαστε στην Πορτογαλία και τον Πέντρο Ντουάρτε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ξεκινήσω ευχαριστώντας άμεσα για την... Ε, εδώ βρίσκομαι γιατί να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τον αναλυτικό τρόπο με τον οποίο ε, μας ε, κάνατε την εισήγησή σας και θέλω να κάνω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη ήδη κατά κάποιο τρόπο αναφέρθηκε στην πρώτη παρέμβαση από τον αυστριακό συνάδελφο και αφορά την κρίση των, του δημόσιου χρέους που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες ε, και που επιδεινώνεται λόγω των διαφόρων πιέσεων, λόγω της συγκυρίας αλλά και λόγω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτά τα επιτόκια λοιπόν που μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι ε, βιώσιμα Εσείς θεωρείτε ότι με βάση αυτόν τον μηχανισμό που είπατε σταθερότητας και που ήδη συμφωνήσατε θα θα βοηθήσει, θα αρκέσει μάλλον για να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση. Αν ε, όμως υπάρξουν άλλου είδους ε, περιστάσεις, όπως ας πούμε μια διακύμαση αυτών των επιτοκίων θα είναι απαραίτητη για να σωθεί η κατάσταση σε ορισμένες χώρες της ε, Ευρώπης και μέσω... με βάση αυτή την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε τώρα για το ευρώ και έπειτα το σύμφωνο ευρώ. Είναι πολύ σημαντικά μέτρα όντως για να δοθεί σταθερότητα και ισχύ στο κοινό μας νόμισμα. Εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι ισορροπία ανάμεσα στον οικονομικό προγραμματισμό, πράγμα που όλοι περασπιζόμαστε, και τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους, το κοινωνικό και οικονομικό του πλαίσιο και κατάσταση. Θεωρείτε δηλαδή ότι εντός αυτού του συμφώνου θα γίνει σεβαστή η ιδιαιτερότητα του κάθε κράτους, θα μπορέσουν να δοθούν διαφοροποιημένες απαντήσεις, οι καλύτερες δηλαδή για κάθε περίπτωση και από την άλλη πλευρά ταυτόχρονα να γίνει σεβαστή η κυριαρχία του κάθε, κάθε κράτους μέλους και η δυνατότητα των ερετών του κάθε κράτους να καθορίζουν τη μακροοικονομική τους πολιτική. Συντονισμός οικονομικός βεβαίως ναι, αλλά οι πληθυσμοί μας να ερμηνεύσουν αυτό το σύμφωνο όχι ως ε, συντονιστικό μέσο, αλλά ως μια απόπειρα επιβολής ε, οικονομικής πολιτικής, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οικονομικοί και κοινωνική και επιπτώσεις αυτού του συμφώνου. Πώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Σας ευχαριστώ. Α, μπορούμε να βγούμε και από την Ευρωζώνη να πάμε στη Ρουμανία. στον κύριο Βοσγανιάν. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του κυρίου Πρόεδρου. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα σημαντικό στάδιο στη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα του προπολογισμού, να, τα, να τον ενισχύσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Ε, το 2010 Φερρυπίν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν διορθωτικές ως, αλλαγές όσον αφορά τα ελλείμματα οδήγησαν σε μείωση την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει ε, επενδύσεις σε δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μέλλον θα έχουμε δυσκολίες να επιτύχουμε αν έχουμε ε, αντιμετωπίζουμε το, την κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο χωρίς να πάρουμε κάποια μέτρα και να κάνουμε μείωση των δαπανών. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, όταν μιλάμε για συντονισμό, Φερρυπίν, συντονισμό στο θέμα των προϋπολογισμών, τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει είναι σαφέ ότι πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένους κοινού στόχους. Υπάρχουν τώρα χώρε όμω που έχουν πολύ διαφορετική κατάσταση όσον αφορά τον προπολογισμό. Ποικίλει από τη μια χώρα στην άλλη. Άλλε χώρε έχουν ε, φέρει πίν ε, έσοδα που είναι υπέ, ε, παραπάνω, δηλαδή πλεόνασμα 300% και άλλε χώρε οι οποίε βρίσκονται σε ένα επίπεδο 30%, άλλε σε ένα χαμηλότερο, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι θα είναι σημαντικό για να, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε ε, να συντονίσουμε μάλλον τις εθνικές οικονομίες, ούτως ώστε να έχουν αυτές οι οικονομίες τις ε, κοινέ προϋποθέσεις για να πετύχουν τους στόχους της ε, στρατηγικής για το 2020. Τώρα, ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την, αυτό που λέγαμε την, ε, αν έχει η Ευρώπη δηλαδή την ικανότητα, την εμπειρογνωματοσύνη, την έχουμε. Φιλιππίνη χώρα μου, ε, στο 2009 είχαμε την πρόγνωση της Επιτροπής, η οποία όμως ήταν λαθεσμένη. Εμείς είχαμε μια μείωση όσον αφορά την εξέλιξη. Είχαμε μια πρόβλεψη φέρει πριν αργότερα του 1,5%, εμείς καταλήξαμε σε 1,2%. Είναι λοιπόν σαφέστατα ότι θα πρέπει να μπούμε πλέον και σε νέους τομείς. Έχουμε να κάνουμε τους τομείς που έχουν να κάνουμε με την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η πρόεδρος. Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να συντομεύετε τι παρεμβάσει γιατί ο πρόεδρο ε, Φανορών Ποϊ πρέπει κάποια στιγμή να φύγει. Και έχω ακόμα τρει που έχουν ε, ζητήσει το λόγο. Πράσινη κάρτα λοιπόν από την ε, Λιθουανία και τον κύριο Τουκάτη. Έπειτα. Είναι Τβέλτ και Πόρτας. Παρακαλώ ε, τους ευρωβουλευτές να τα πούν σε ένα λεπτό που είναι συνηθισμένοι. Gerai, Μάλιστα. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Φάνο Ρομπόη που είσαστε εδώ μαζί μας και παρουσιάζετε αυτές τις ιδέες. Είναι κρίμα ότι στη Λιθουανία δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή να υπάρξει μια συζήτηση αυτό εδώ το θέμα. Συμφωνούμε όμως όσον αφορά την ε, ειδικό, ιδιαιτερότητα που υπάρχει όταν έχουμε να κάνουμε 27 χώρε, Έχουμε θέματα τραπεζικής φύσεως. Φέρει πίν στη Λιθουανία, ξέρετε. Έχουμε... Έχουμε το μοντέλο που έχει να κάνει με σταθερό ε, ε επιτόκιο όσον αφορά τις συναλλαγές. Θα ήθελα να ξέρω, θα δημιουργήσετε μηχανισμούς οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τα ισχύοντα οικονομικά και κοινωνικά μοντέλα. Θα το λάβετε αυτό υπόψη. Και επίση όσον αφορά τις σταθερές, ε, τα σταθερά επιτόκια συναλλαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον ε, κύριο Φαναρομπόη. Καλωσορίζω τους εθνικούς συναδέλφους. Είμαι πολύ ευτυχής που τόσοι πολλοί ήρθατε θα πρέπει να πω ότι αφού είδα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας και τις συζητήσεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη και ανήσυχη. Διότι για να είμαι ειλικρινή, θα πρέπει να σα πω ότι τα έχουμε ξανακούσει τα ίδια. Λέτε πω το ευρώ είναι σταθερό, αλλά το ευρώ είναι τόσο σταθερό όσο και η πολιτική βούληση που το στηρίζει. Και αυτό και η πολιτική βούληση τελευταία φαίνεται να είναι πολύ μικρή. Γιατί αδύναμη, γιατί δεν καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε την αυστηρά διακυβερνητική προσέγγιση. Ε, Πάντα στου επισκέπτε μου που έρχονται εδώ, του λέω, αν είναι μια ομάδα 27 ανθρώπων, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα του δώσει ε, σάντουιτς με τυρί ή με, με ζαμπόν. Άμα χρησιμοποιούσαμε την ομοφωνία, μάλλον θα μένανε όλοι νηστικοί. Φανταστείτε για κάτι πιο περίπλοκο. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Και ακριβώ αυτό συμβαίνει. Η Ευρώπη έχει τελματώσει και μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε και να συζητάμε από μακρόν για τα πιο φάρμακα χρειάζονται. Αλλά άμα ο άρρωστος δεν θέλει να καταπιεί το χαπάκι, μπορούμε να συζητάμε ή θα παραμείνει άρρωστος. Ο υπόλοιπο κόσμο όμω δεν περιμένει εμά. Ναι, Πρόεδρε, βλέπω που μου κάνετε νόημα να κλείσω, γιατί έχω μια πολύ απλή ερώτηση που περισσότερο έχει σχέση, με, ε, μάλλον την απευθύνω προς ε, συναδέλφους εδώ, και, αλλά την απευθύνω και σε εσά. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουν τα κράτη-μέλη. Το όχι, ξέρω να το λένε πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι επιθυμούν, όχι μόνο για το κράτος μέλους τους, αλλά για την Ευρωζώνη. Γιατί αν τα κράτη-μέλη δεν αναλάβουν την ευθύνη για την Ευρωζώνη και την Ευρώπη γενικότερα, τίποτα δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μιγκουέλ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φανορμπόη, η κυβέρνηση της χώρας μου, της Πορτογαλίας, έδωσε την τελευταία Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το τέταρτο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Το έγγραφο αυτό δεν συζητήθηκε με κανέναν εταίρο, δεν συζητήθηκε με κανένα κόμμα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και ο κύριε Πορομπόη έρχεστε εδώ και μου λέτε πως ο ρόλος των εθνικών βουλευτών στον οικονομικό συντονισμό είναι πολύ σημαντικός. Μα τελικά τι να πιστέψουμε, τα λόγια σας ή την πράξη των, της κυβέρνησης. Δεύτερη ερώτηση. Υπολογισμό του ελλείμματος. Οι Γερμανοί στις αρχές του ευρώ είχαν μια θεμητή άποψη σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες επενδύσεις θα έπρεπε να αφαιθούν εκτός του υπολογισμού του ελλείμματος. Τουλάχιστον οι επενδύσεις για το σχηματισμό του σταθερού κεφαλαίου ερώτησή μου είναι, γιατί στον υπολογισμό του ελλείμματος δεν υπερασπίζεται το Συμβούλιο ότι τα επιτόκια του ελλείμματος να βρίσκονται απ' έξω, δηλαδή το έλλειμμα να υπολογίζεται ως κύριο, ε, πρωτογενές μάλλον ε, υπόλοιπο, πράγμα το οποίο θα επέτρεπε να υπερασπιστούμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν τις περισσότερε δυσκολίε, που όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, χωρίς να μπορούν να αναπτυχθούν, μπορούν όμως να μειώσουν το έλλειμμα αλλά δεν, κατα... το... αλλά δεν ε, καταφέρουν να μειώσουν το χρέος, γιατί αυτή είναι η πολιτική, εκεί μας οδηγεί η πολιτική που ακολουθείτε. Τελευταία μου ερώτηση είναι πώς θέλετε να πείσετε τις χώρες να καταφύγουν στο Ταμείο Σταθεροποίησης αφού είναι δάνεια με 6% όπως αυτά που δόθηκαν στην Ιρλανδία και τελικά ε, επηρεάζουν τους μισθούς αλλά δεν αγγίζουν τη φορολογία. Γιατί δηλαδή, με άλλα λόγια, ε, να πληρώνουν πάντα οι ίδιοι. Thank you. I think... Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα περισσότερα ήταν σχόλια παρά ερωτήσεις. Ε, κύριε Πρόεδρε, κάντε ό,τι μπορείτε σε τόσο λίγο χρόνο που έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρεμβάσεις στα γαλλικά παρόλο που θα πρέπει να απαντήσω πολύ σύντομα, αλλά πραγματικά με προβληματίζουν. Καταρχήν, μία παρατήρηση. Όσοι προσάπτουν στην Ευρώπη ή στα θεσμικά της όργανα ότι είναι αργά, ότι δεν είναι δυναμικά, αδρούν ίσως καθυστερημένα, υπενθυμίζω όταν άρχισα, ανέλαβα αυτό το αξίωμα δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα σύμφωνο σταθερότητα το οποίο δεν εφαρμόζεται. Δεν υπήρχε κανένας μακροοικονομικός έλεγχο. Τίποτα. Τίποτα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ούτε για τη φούσκα την, ε, την κτηματιστηριακή. Ε, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και δεν υπήρχαν ταμεία διάσωση. Τίποτα. Ούτε περιστασιακά, ούτε προσωρινά, ούτε... Τίποτα δεν υπήρχε. Λοιπόν, όταν πρέπει κανείς να δράσει όπως και έπρεπε είναι διότι δεν υπήρχε τίποτα προηγούμενο. Αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση. Διότι πολλοί μας ασκούν κριτική πολύ εύκολα. Χρειάστηκε ε, δηλαδή να ληφθούν κάποια μέτρα. Θα πρέπει απ' την άλλη να αποφύγουμε ούτως ώστε αυτή η οικονομική κρίση να ξαναεπαναληφθεί. Γι' αυτό και πήραμε κάποια διαρθρωτικά μέτρα Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, είναι οι έξι προτάσεις της Επιτροπής, είναι η έκθεση για την, ε, της Task Force και σήμερα προσθέσαμε το σύμφωνο για το ευρώ. Είναι διαρθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη διακυβέρνηση, ούτως ώστε αυτή η κρίση να μην ξαναεπαναληφθεί στο μέλλον. Λοιπόν, είναι βασικό στοιχείο αυτό Τώρα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα είναι μόνιμος όσον αφορά τις κρίσεις μετά το 2013. Έχουμε λοιπόν την οικονομική διακυβέρνηση και τις παρεμβάσεις οικονομικές όσον αφορά για την διάσωση. Υπάρχουν δηλαδή πρωτοβουλίες οι οποίες, ε, οι οποίες θα λέγαμε είναι τέτοιες για να μπορέσει κανείς στο μέλλον να ελέγχει τις κρίσεις. Στο μέλλον λοιπόν θέλουμε να αποφύγουμε μια κρίση και αυτό είναι το βασικότερο. Τρίτη παρατήρηση. Μήπως τα μέτρα που έχουν λήφθει θα αρκούν για να σταθεροποιηθεί η κρίση στην Ευρωζώνη. Όχι για το ευρώ, γιατί το ευρώ είναι ισχυρό νόμισμα. Και τώρα, μήπως κάποιες χώρες που παίρνουν μέτρα ε, θα μπορέσουν να τα καταφέρουν αυτά τα μέτρα. Εγώ Στη χώρα μου ήμουν υπουργό οικονομικών. Όταν είχαμε να κάνουμε την ε, κρίση ε, για τον προπολογισμό, όπου είχαμε ένα, ε, ένα ποσοστό του 130% του ΑΕΠ. Και μας δόθηκε τότε ο χρόνος, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, μας δόθηκε ο χρόνος στη δεκαετία του, του 90, ακόμα και του 80, αλλά κυρίως του 90, είχαμε το χρόνο να ε, να πάρουμε μέτρα, διαρθρώσουμε, ούτω ώστε να μην, τα δημοσιονομικά μας να μην αποτελούν πρόβλημα. Ο Υπουργό τη Σουηδία, στην τελευταία συμβούλιο στην Ευρώπη, μα είπε: Είχαμε μια κρίση στη Σκανδιναβία τώρα, τέλη τη δεκαετία 80, αρχέ 90. Είχαμε λοιπόν μια κρίση δημοσιονομική και οικονομική και μας Είχαμε στη διάθεσή μα 8 χρόνια για να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Και τα καταφέρουμε, όπω και στη χώρα μου εξάλλου. Λοιπόν, άρα χρειάζεται χρόνο. Και φυσικά, αυτό είναι το νέο στοιχείο για την δημοσιονομική αγορά. Δηλαδή, η, η, για τις χρηματαγορές, συγγνώμη. Στα πρώτα δέκα χρόνια της ιστορίας του ευρώ δεν υπήρξε αντίδραση. Σήμερα αντιδρούμε στα πάντα. Με το παραμικρό υπάρχει ε, υπερβολική αντίδραση. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή και ο Επιτροπός Μπαρνιέ πήραν μια σειρά μέτρων, δημιουργήσαν μια πανοπλία θα λέμε, μια μεγάλη πρωτοβουλία, πολλές μάλλον, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ε, διορθώσουμε, να ελέγξουμε καλύτερα τις ε, ε, αγορές. Επίση, έγινε μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο έλεγχο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό, θα έλεγα. Ούτω ώστε να ε, αντιμετωπιστούν όλε οι κερδοσκοπικέ τάσει και να ε, προβλεφθούν ορισμένε υπερβολέ όσον αφορά τα δημοσιονομικά θεσμικά όργανα. Τώρα, φυσικά, όμως μπροστά μα έχουμε μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την σταθεροποίηση των δημοσιονομικών. Αυτό είναι απαραίτητο και αναπόφευκτο και για τις ε, εθνικές πολιτικές, διότι ε, έχουμε την Ευρωζώνη, θέλουμε να εξηγιανθούν τα δημοσιονομικά, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ένα καθήκον ε, εθνικό θα λέγαμε. Η Ευρώπη φυσικά και σκουντάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σε σε εθνικό επίπεδο, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί ε, μελλοντικά ε, το, δικό μας κοινωνικό μοντέλο. Στα πλαίσια όμως αυτής της ε, δημοσιονομικής ε, ε, προσπάθειας θα πρέπει να δούμε την ανάπτυξη για το μέλλον, την κατάρτιση και άλλες πτυχές και αυτό, αυτά θα λέγαμε ότι αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε εδώ το ευρωπαϊκό εξάμεινο υπάρχει ένας έλεγχος πολύ συγκεκριμένο, όχι μόνο για την ε, σταθεροποίηση, εξυγίανση των, ε, των δημοσιονομικών και τα, μακροοικονομική, αλλά να δούμε και τη στρατηγική του 2020, η οποία θα πρέπει να ενωσοματηθεί σε αυτές τις άλλες προσπάθειες. Να μην γίνεται μια μονομερής ανάπτυξη για μια, ας το πούμε, δημοσιονομική πειθαρχία ή Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο μόνο του, να μην το αφήσουμε να εκφυλιστεί θα λέγαμε σε μια γραφειοκρατική διαδικασία, να το πάρουμε στα σοβαρά και τις τρεις συνιστώσεις αυτού και να αναπτυχθούμε προς μια οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλοί από εσά ε, και με το δίκαιο του, ε, επιμείναν σε αυτό που έχει να κάνει με τις παραδόσεις σε κάθε χώρα για να εφαρμόσουμε τους κοινούς αυτούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν, από την αρχή εγώ απέρριψα ορισμένα έγγραφα που κυκλοφορούσαν στον τύπο, Φερρυπίν, όσον αφορά τις συντάξεις, τα συστήματα, ε, όσον αφορά το όριο ηλικίας συνταξιότητας 67 ετών, και διάφορα συστήματα που ισχύουν στις χώρες. Αυτή δεν είναι η σωστή μέθοδος. Το θέμα της αυτόματης συμμετοχλητικής ε, Εδώ έχουμε να κάνουμε με αρμοδιότητες που είναι σε εθνικό επίπεδο. Εθνικά κοινοβούλια θα πάρουν τις αποφάσεις. Έχουμε φυσικά άλλα όργανα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα που θα έχει σαν στόχο να ελέγξει αν οι στόχοι επιτευχθεί και ο τρόπος με τον οποίο έχουν επιτευχθεί. Αλλά ε, καταρχήν έχουμε τις ευθύνες σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμός, έλεγχος, ενδεχομένως κάποιες κυρώσεις. Υπάρχει φυσικά και η πίεση της αγοράς, υπάρχουν η πίεση από τα θεσμικά όργανα. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος η αρμοδιότητα είναι σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε φυσικά ε, υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με ε, επικαλύψεις και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ότι πολλά στοιχεία του συμφώνου θα πρέπει να ενταχθούν, να σωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το έχουμε προβλέψει. Αλλά θέλουμε να, να ασκήσουμε λίγο μεγαλύτερη πίεση, πέρα από την πίεση που υπάρχει. Γι' αυτό άπαξε τη στο μεγαλύτερο ε, σε υψηλό επίπεδο με όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία συντονισμού. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν άπαξ ε, του έτους με, με βάση τη σύσταση Επιτροπής να δώσουμε μια περαιτέρω πίεση αν χρειαστεί. Διότι έχουμε ένα κοινό νόμισμα και θα πρέπει να έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία πάει προς στην ίδια κατεύθυνση και θα πρέπει μια οικονομική πολιτική η οποία μπορεί να μην είναι ταυτόσιμη αλλά πάει προς την ίδια κατεύθυνση. Θα αρκέσουν όλα αυτά. Ο μηχανισμός για την, ε, ο μηχανισμός επέμβασης θα αρκεί. Δεν ξέρω, να είμαστε ρεαλιστές. Ο μηχανισμός που έχουμε σήμερα είναι ένας που χρησιμοποιήθηκε για 17 δις 250 εκατομμύρια είναι ήδη διαθέσιμα και 240 θα χρησιμοποιηθούν αφού το εφαρμόσουμε το σύμφωνο. Το πρόβλημα δεν είναι εδώ. Θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά την οικονομία σε ορισμένες χώρες και αν υπάρξει ανάγκη είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε. Είμαστε έτοιμοι για την Ελλάδα. Δεν υπήρξε κάτι που είχε προβλεφθεί πριν, όπως ξέρετε, στο σύμφωνο της ε, Λισαβόνας. Τίποτα δεν είχε προβλεφθεί τα πρώτα δέκα χρόνια και το κάναμε τώρα. Και θα κάνουμε τα πάντα για να σταθεροποιήσουμε την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Τα πάντα. Και τότε δεν θα λείψουν τα μέσα. Και τελευταία παρατήρηση. Μερικοί από εσά παραπονέθηκαν και δικαιολογημένα όσον αφορά τα μέτρα λιτότητος. Θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, ε, με δίκαιο ε, στα πλαίσια μιας χώρας. Είναι σημαντικό αυτό από την κοινωνική πτυχή και αυτή η πτυχή είναι, είναι Εγώ φέρει είμαι από μια χώρα η οποία αρχές του, τη δεκαετία του 80 ξεκίνησε με ένα έλλειμμα 15%. Δεν το συγκρίνουμε με το ελληνικό. Εμείς πετύχαμε με, με διάφορους ε, προσπάθειες, ε, να έχουμε μια, κοινωνικές, ε, μια κοινωνική προσέγγιση η οποία μας οδήγησε έξω από την κρίση. Με διάφορες συμμαχίες το πετύχαμε αυτό. Σήμερα, λοιπόν, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ε, το, αυτό που κάνουμε σήμερα να είμαστε σίγουροι για το μέλλον. Δεν είμαστε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την πτυχή που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και την κοινωνική πτυχή. Και πούμε στους ανθρώπους, στον κόσμο, ότι είναι μια προσπάθεια, μια προσπάθεια, ε, παρόλο που είναι δύσκολη, και ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιες χώρες υποφέρουν σήμερα. Αλλά αυτό τι, τι, στόχο έχει. Όχι να καταστρέψουμε το οικονομικό μας μοντέλο, αλλά να το διασώσουμε. Είναι προσπάθειες, είναι ούτω ώστε στο τέλος να κερδίσουμε τη μάχη όσον αφορά το δικό μας κοινωνικό μοντέλο. Και όχι να το καταδαφίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων υπάρχει μια εθνική ευθύνη. Εμείς δίνουμε τους στόχους, τους διασαφηνίζουμε, τους μεγάλους στόχους, οικονομική, όσον αφορά τον προπολογισμό, διαρθρωτικές αλλαγές, αλλά όσον αφορά την εφαρμογή, αυτό είναι ένα θέμα που εντάσσεται στην εθνική ε, αρμοδιότητα. Φυσικά έχουμε την, την ευρωπαϊκή μέθοδο η οποία μας επιτρέπει να ασκούμε πίεση και αυτοί που δεν, ε, δεν εντάσσονται σε αυτή την πειθαρχία, ε, τότε, σε τέλος, τέλος, τέλος, μπορεί να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις, ούτως ώστε όλοι, μα όλοι, να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντοτε σεβόμενοι τις εθνικές αρμοδιότητες. Αυτά σαν αντιδράσεις όσον αφορά τις παρατηρήσεις που κάνατε, οι οποίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες Ουσιώδης, Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ξέρω ότι πρέπει να φύγετε αμέσως. Ελπίζω να μην σας καθυστερήσαμε και χάσετε το αεροπλάνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα ε, Δώσω λίγων λεπτών. Λοιπόν, μην παραχαλαρώσετε, γιατί θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε αμέσω στην επόμενη ενότητα. Λοιπόν, περνούμε στο επόμενο θέμα της ημέρας της διάταξης που είναι ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε ένα πάνελ τεσσάρων Προέδρων Επιτροπών. Από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ο κύριος Κλάινα, ο κύριος Βάνμπρουκ, ο κύριος Καζουάκ και ο κύριος Στουμφόλ. Και τέσσερις είναι συγητές ε, ε, της δέσμης μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης. Παρακαλώ, όσοι εξέρχεστε τις αιθούσεις θα το πράξετε ησύχως, γιατί θα χάσουμε και άλλο χρόνο. Τώρα, πώς έχει το χρονοδιάγραμμα. Κάθε ένας από τους πάνελις θα μιλήσει για πέντε λεπτά και μετά ερωτήσεις να σας θυμίσω ότι αν θέλετε για αυτή την ενότητα να ζητήσετε το λόγο, σηκώνετε τη γαλάζια κάρτα. Σας παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία. Ε, μιλάτε όσο μιλάω εγώ, αλλά δεν θα σας αφήσω να μιλήσετε την ώρα που θα ακούμε τους ομιλητές μας. Ε, ο κύριος Κλάινα, πρόεδρος Επιτροπής Προπολογισμού και Οικονομικών της Πολωνικής Γερουσίας. Παρακαλώ. και κύριοι, Μόλις παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή του κυρίου Φαναρομπάη. Η συζήτηση αυτή μας οδήγησε σε ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον που αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η συζήτησή μας εντάσσεται στον κύκλο διακοινοβουλευτικών συζητήσεων που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε πως τα θέματα που θίγουμε μπαίνουν σε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω πως είναι κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε τι πετύχαμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από το μέλλον. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ε, η οικονομική κρίση που ξέσπασε το Σεπτέμβριο 2008 μετά από την κατάρρευση της Lehman Brothers ε, συνεχίζεται. Ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι που βλέπουν τα πρώτα μηνύματα ανάπτυξης ε, γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτή η ανάπτυξη είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Νομίζω πως θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα τελευταία στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020, αλλά να λάβουμε υπόψη και τους περιορισμούς ε, που υπάρχουν ε, για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ρηξικέλευτες και χρειάζονται επίσης ε, πολύ θαραλές αποφάσεις όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέσα. Έχουμε στόχους για το μέλλον. Είναι πρόκειται κυρίως για την ανάπτυξη και τον περιορισμό της ανεργίας. Άρα προφανώς η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν ένα φιάσκο. Και θα πρέπει να έχουμε ένα γενικότερο όρομα για να μπορέσουμε να αντισταθούμε στον ανταγωνισμό που μας έρχεται από την ΣΥΠΑ, από την Κίνα και από άλλες τρίτες χώρες. Έχουμε το πρόγραμμά μας, το Γαλιλαίο, το ΙΤΕΡ κτλ. Αλλά πώς μπορούμε να υποφεληθούμε ώστε να γίνουμε όλο και πιο ανταγωνιστικοί. Χρειαζόμαστε μέσα που μας λείπουν πολύ συχνά όλα δείχνουν πως ο προπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2014 με 2020 δεν θα είναι κατάλληλος σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Έχουμε αμφιβολίες λοιπόν όσον αφορά την υλοποίηση των οικονομικών πολιτικών στα κράτη-μέλη μετά από τις συστάσεις που μας ε, έρχονται από την Κομισιόν. Γίνεται λόγος για την σταθεροποίηση της οικονομίας, για την καταπολέμηση της φτώχειας και νομίζω πως αυτά είναι δύσκολο να συμφιλειωθούν ακόμα και όταν μιλά κανείς με την ε, σημείο εκκίνησης λέγοντας ότι η Ευρώπη η στρατηγική 2020 είναι η μια στρατηγική με μήνυμο στόχους, βλέπουμε πως τα κράτη-μέλη, ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι στόχοι, δύσκολα μπορούν να επιτευχθούν. Μπορεί κανείς να ονειρεύεται βέβαια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κτλ. Αλλά απλούστατα το κονδύλι για την έρευνα και την ανάπτυξη δεν φτάνει παρά μόνο στο 3% το προϋπολογισμό. Η γεωργική πολιτική και η πολιτική σύγκληση είναι απαραίτητες θα πρέπει να μειωθούν οι αποκλήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη και νομίζω πως ο μέσος όρος της Ένωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ακόμα κι αν πάρουμε άλλους δείκτες στα κράτη-μέλη, αν δούμε δηλαδή την ανάπτυξη του ΑΕΠ στις χώρες μέλη, οι αποκλήσεις μπορεί να αυξηθούν κι άλλο. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι υπέρ της πολιτικής σύγκλησης. Είναι κάτι απαραίτητο. για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολυδιάστατη αλληλεγγύη σε επίπεδο ένωσης. Δεν πρόκειται για αλτρουισμό, πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως ένωση. Ποια είναι τώρα τα νέα μέσα διακυβέρνησης σε οικονομικό επίπεδο νομίζω πως γίνεται κυρίως λόγος για την εποπτεία και την, τους νέους θεσμούς. Εγώ νομίζω πως Ίσως είναι υπερβολική αντίδραση σε επίπεδο της Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν νέες απαιτήσει, ναι. Αλλά αυτές οι νέες απαιτήσει δεν αποτελούν τροχοπέδι για τον ανταγωνισμό. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αμφισβητείται αυτό το 3% του ελλείμματος που επιτρέπεται. Ακολουθώντας αυτά τα οποία υποστηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσαμε ίσως να δράσουμε πιο ενεργά για να σώσουμε ορισμένους τομείς. Χώρες όπως η Πολωνία που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη είναι υποχρεωμένες να προχωρούν σε κάποια λιτότητα. Πρέπει να μειώσουμε το έλλειμμά μας και τον δημόσιο προπολογισμό μας. Το κάνουμε, αλλά αυτό σημαίνει ένα σωρό περιορισμούς για μας. Ε, όσον αφορά την Πολωνία, το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιονομικών δαπανών μας είναι σταθερές δαπάνες. Ε, πρέπει δηλαδή να προχωρήσουμε σε περικοπές όσον αφορά την παιδεία, για παράδειγμα, ή την έρευνα. Αυτοί οι δημοσιονομικοί περιορισμοί λοιπόν σε κράτη-μέλη αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε πως η δημοσιονομική πειθαρχία και η λιτότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ταυτόχρονα θα ήθελα να αναφέρω κάποια παραδείγματα, όπως ε, δηλαδή η Πολωνία που μαζί με άλλα νέα, ε, νέα κράτη-μέλη πέρσι ζήτησαν να υπάρξουν ε, μόνιμες λύσεις ώστε η μετάβαση προς τη χρηματοδότηση των συνταξιδοτικών ταμείων να μην ληφθεί υπόψη. Είδαμε όμως πως αυτό δεν έγινε δεκτό. Δηλαδή, κάθε κράτος βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση οικονομική και δημοσιονομική και θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ανεξάρτητα τώρα από αυτά που είπα, βλέπουμε θετικά τις διάφορες πρωτοβουλίες όσον αφορά το συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών στα κράτη-μέλη και ελπίζουμε πως το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο. Τώρα όσον αφορά τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις ε, κυβερνήσεις ε, γίνεται τακτικά. Ε, είμαστε τώρα στην αρχή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και δεν θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες υπερβολικά αυστηροί σε αυτό το επίπεδο, διότι τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο θα ήταν πρόημο κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν πως ε, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συνεργασίας είναι αυτά που θα μετρήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Διευκρινιστικά ε, πρέπει να σας πω ε, ότι στην αρχή είχαμε δώσει 7 λεπτά στους ηγητές μας και τώρα τα κάναμε 5 και τους δυσκολεύουμε, τους περιορίζουμε. Κύριος Βαντιμπρούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις είπα και προηγουμένως στο Βελγικό Κοινοβούλιο κάναμε εκτενέστατη συζήτηση μετά από ερωτήσεις που μας είχαν στείλει. Αρχικά ήταν ε, καινούργια η διαδικασία αυτή για μας. Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμη. Ήταν ευρύτατη η συνένεση την οποία πετύχαμε όλα τα δημοκρατικά κόμματα για μια απάντηση έτσι αρκετά ουσιαστική και περιεκτική. Τόνισα ήδη στη συζήτηση ένα στοιχείο, θα ήθελα να το επαναλάβω και να προσθέσω και μερικά ακόμα επιγραμματικά. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε εμείς ότι είναι πολύ σημαντικό το ευρωπαϊκό εξάμεινο και η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να εγγράφεται σε μια στρατηγική που να στρέφεται προς την οικονομική ανάπτυξη και να είναι αρκετά ευρεία όσο και ισορροπημένη. Επίσης θεωρούμε ότι το στοιχείο της πρόληψης νέων ε, οικονομικών και χρηματοοικονομικών κρίσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πρώτα σε αυτό το τελευταίο, την πρόληψη. Έχουμε την αίσθηση στο Βελγικό Κοινοβούλιο ότι ορισμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συζήτηση ε, για το χρηματοοικονομικό τομέα σήμερα τείνουν να μας διαφεύγουν στην Ευρώπη. Δεν τα προσέχουμε, δεν τα σκεφτόμαστε. Ας πούμε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των τραπεζών που είναι τράπεζες για αποταμίευση, για καταθέσεις και κάποιες άλλες τράπεζες που είναι τράπεζες εμπορικές με μεγαλύτερο ρίζικο. Και ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, αυτό γίνεται, αυτή η διάκριση όλο και περισσότερο. Στην Ευρώπη όχι. Εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι λοιπόν να κάνουμε ε, μία διάκριση μεταξύ των ε, παλαιών κλασικών ε, τραπεζών για τις καταθέσεις και των εμπορικών πιο επιθετικών τραπεζών. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε άλλα μέτρα. Βασιλεία 3. Είναι μια λέξη κλειδί, ε, επίκυνται αυτές οι συμφωνίες ε, και ε, είναι επίσης το θέμα της διαθήκης των τραπεζών όταν συνδυάζουν ε, τις ε, κλασικές καταθετικές ε, δραστηριότητες με τις πιο επιθετικές από πλευράς τραπεζών, πιο εμπορικές. Ξέρω ότι θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα της Βασιλείας 3 και θα παρακαλούσαμε να ληφθούν υπόψη και αυτά τα διαρθρωτικά ζητήματα του τραπεζικού τομέα και του τραπεζικού τοπίου όπως το λέμε. Και χρειάζονται λοιπόν διαρθρωτικές αλλαγές ε, στο τραπεζικό τοπίο στην Ευρώπη και θα τα δει αυτά η βασιλιατρία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μας έχουν ξεπεράσει, παίρνουν ε, αποφάσεις σημαντικέ ε, πιο γρήγορα από ότι η Ευρώπη. Έρχομαι τώρα στην τόνωση τη οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης τη οικονομία. Λέμε στην έκθεσή μας ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε την ενοποίηση τη Ευρωπαϊκή εσωτερική Αγορά και παραπέμπουμε στην έκθεση Μόντι, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη συγκεκριμένα. Γνωρίζω ότι αυτό το θέμα είναι κάπως επίμαχο, αλλά στο Βελγικό Κοινοβούλιο είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία υπέρ ε, της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, των διασυνοριακών μεγάλων έργων με ευρωομόλογα, αυτά τα project bounds ε, ομόλογα. τα ομόλογα δεν αφαιρούν την ευθύνη από τα κράτη-μέλη. μπορούν να παίξουν το ρόλο τους και μπορούμε να αναπτύξουμε και νέα μέσα και εργαλεία χρηματοδότησης στον χρηματοοικονομικό τομέα και εδώ παραπέμπουμε ε, στο φόρο ή στο τέλος ε, χρηματικών, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επίση, είπα και προηγουμένω, θεωρούμε ότι οι συμφωνίες που θα προκύψουν θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά, αυστηρά στην πράξη. Αλλά με ένα ευρύτερο όραμα για το τι ε, θα προωθεί στην Ευρώπη προς τη στρατηγική 2020. Μια απαραίτητη στρατηγική ανάπτυξης. Αυτό βλέπουμε και στον τόνο που δίνεται και ε, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, αλλά όχι μόνο σε αυτό, και στην παιδεία, ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να ε, δούμε και κάποια άλλα θέματα κοινωνικά, κοινωνική συμπερίληψη, απασχόληση, ποιότητα της εργασίας. Για να είναι η Ευρώπη αξιόπιστη θα είναι σημαντικό όταν κάνουμε λοιπόν συστάσεις στα κράτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ε, Οικονομικής Διακυβέρνησης για το 2020, αυτές οι συστάσεις δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τη δημοσιονομική πειθαρχία, ούτε αποκλειστικά ε, την ανταγωνιστικότητα, αλλά θα πρέπει να αναφέρονται και στην έρευνα, στην ανάπτυξη, στις προσπάθειες που πρέπει να γίνονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην κοινωνική συμπερίληψη. Αυτά, Πρόεδρε γιατί δεν έχω και άλλο χρόνο, ορισμένα στοιχεία από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Thank you very much. Uh, next... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο κύριος Καχούζακ και ζητώ συγγνώμη για το τυπογραφικό σφάλμα στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που καλέσατε τους εθνικούς βουλευτές και τους συνδέσατε με τις εργασίες σας. Πιστεύω πως η συνεργασία αυτού του τύπου είναι απολύτως απαραίτητη. Είναι αλήθεια πως ο καθένας έχει να παίξει έναν ρόλο εφόσον είναι νόμα εκλεγμένος. Φυσικά και τα θεσμικά όργανα ταλανίζονται από την κρίση του δημόσιου χρέους που γνωρίζει ο ολόκληρη Ευρώπη, αλλά λύσει που να είναι σκόπιμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρί την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ μας ε, για ε, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Να σας πω δύο λόγια για το πώς εμείς προβλέπουμε στη Γαλλία το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μετά θα αναφερθώ και στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Μέχρι το 2010 το, η γαλλική κυβέρνηση διαβίβαζε στο κοινοβούλιο ότι ο περιεχόμενο των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει πριν, αφού το είχε παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέταση το, των μεταρρυθμίσεων, άρα λοιπόν εκ των προτέρων δεν είχε λόγο λοιπόν ε, ύπαρξη στη φάση τη συζήτηση στο Εθνικό Συνέλευση, αφού ούτως ή άλλω είχε διαβιβαστεί αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε υποθέσει και στόχους του οποίων θα πρέπει να γίνει μετάφραση στον εθνικό προπολογισμό. Άρα αυτό το περιεχόμενο θα μπορούσε να, σημειώσει, να χρησιμεύσει ως σημείο σύγκριση για να δούμε τι είχε γίνει ε, για μας του Ευρωβουλευτές. Τώρα, από πέρυσι η, η γαλλική κυβέρνηση προβλέπει και εξετάζει ένα πρόγραμμα τριετές, επεμπνέεται από το ίδιο το πρόγραμμα σταθερότητας, χωρίς να συγχαίει με αυτό όμως. Δύο προγράμματα υιοθετήθηκαν, το ένα το 2009 που βεβαίως ε, ε, ε, δεν στάθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης και ένα άλλο υποβλήθηκε για το 2011 με 2014. Ε, η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει στο Εθνοσυνέλευση το πρόγραμμα αυτό 15 μέρες τουλάχιστον πριν το υποβάλει στα κοινοτικά όργανα. Και έτσι το Εθνικό Κοινοβούλιο νομίζουμε πως ε, συνδέεται πολύ περισσότερο με τα όσα κάνει η γαλλική κυβέρνηση με τους εταίρους της ε, στο πλαίσιο των κοινοτικών θεσμικών όργων. Πιστεύουμε θα πρέπει να παραλαμβάνουμε παρέμβουμε πάντα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την, με, ένα σημαντικό, σημαντικό ψήφισμα για, μέσα σε ένα σύστημα διάδρασης ε, με το Εθνικό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όμως ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για ένα πρόγραμμα σταθερότητας σαν αυτό να ήταν αποκομμένο από την υπόλοιπη οικονομία και απο, αποκομμένο από την επιρροή των διεθνών αγορών. Απαραίτητο λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο να συνδεθούν με αυτή τη διαδικασία. Αλλά πώς, κανένα κοινοβούλιο δεν θέλει να εγκαταλείψει την δημοσιονομική του κυριαρχία και να δώσει δικαίωμα ακόμα και ε, διαβούλευσης για τον εθνικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, ε, θα πρέπει στο πλαίσιο της κυβέρνησής του να εκφράσει ο καθένας ε, τις παρατηρήσεις του. Αλλά αυτό θα μας έκανε να χάσουμε χρόνο. στόχος λοιπόν για τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων θα έπρεπε να είναι μια ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών. Όχι να γίνει μια συνάντηση όπου κάποιοι θα δίνουν διδάγματα στις χώρες τις πιο αδύναμες, αλλά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάποιε εθνικέ ιδιαιτερότητε. Και ορισμένοι συνάδελφοι που εκφράστηκαν πριν από μένα ε, ξέφρασαν την ίδια άποψη και συμφωνώ μαζί του. Πιο συγκεκριμένα οι πρόεδροι των Επιτροπών Προπολογισμού των κρατών μελών θα μπορούσαν να συναντηθούν νωρί μέσα στον χρόνο από τη στιγμή που θα είναι γνωστές, γνωστοί βασικοί ανατολισμοί και πριν από τη θέσπιση του προγράμματο σταθερότητας ώστε να μπει αυτό στην ημερήσια διέταξη και να γίνει έτσι μια ανταλλαγή απόψεων που θα διεύρυνε τη συζήτηση και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάποιε παρατηρήσει, αν μου επιτρέπετε, αν και ήδη έχω μάλλον ξεπεράσει το χρόνο ομιλία, θα ήθελα να εγκρίνω προσωπικά βεβαίω τη μέθοδο του κ. Γαναρομπόη για το σύμφωνο που, στόχο, που θέτει ένα στόχο, αλλά δεν δεσμεύει για τη μέθοδο επίτευξή του. Ε, κάθε κράτο βεβαίω θα πρέπει να επιτύχει του στόχου του. Θα ήθελα να πω ότι η πρόσφατη απόφαση για νομισματοποίηση τουλάχιστον ενό μέρου του, του κυρίαρχου χρέου, του δημόσιου χρέου κάποιων κρατών είναι κάτι το καλό που θα μπορούσε να επιτύχει επιτρέψει να αποφευχθεί επιδείνωση μέσω των κερδοσκοπικών φαινομένων της κρίσης του δημόσιου χρέου κάποιων κρατών και έτσι Χαίρομαι που ορισμένα οι εθνικοί βουλευτές θέλουν να θεσπιστεί ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και μάλιστα ορισμένα κοινοβούλια μπόρεσαν να υιοθετήσουν απαγόρευση για τις ακάλυπτες πωλήσει εγγυήσεων που συνδέονται με τα, τους τίτλους δημόσιου χρέους. Τουλάχιστον είναι μια απόφαση ε, που πλειοψηφική ώστε να μην επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κρίση του δημόσιου χρέου, που ήδη είναι πολύ δύσκολη. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε χρόνο και συγγνώμη που το ξεπέρασα. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν ξεπεράσατε κατά πολύ τον χρόνο σας. Ο κύριος Στομφόλ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της κοινή συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, συμφωνώ πολύ με τον πρόεδρο Φαν Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όλο και περισσότερο ε, σημαντική αυτή η συνεργασία. Και πολλά από αυτά τα πράγματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι στα χέρια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα να το πάω και ακόμα παραπέρα εγώ και να πω ότι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 θα επιτύχει τότε και μόνο τότε εάν τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να εφαρμόσουν τους στόχους τη στρατηγική, να τα εντάξουν στα εθνικά τους προγράμματα και αντίστοιχα να πράξουν. Σε ό,τι αφορά την Αυστρία, εμείς στενιζόμαστε πλήρως αυτό το στρατηγικό τρίγωνο όπως ονομάζεται ε, για ε, την εξηγίαση δηλαδή του προπολογισμού, ε, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Αυτά τα τρία είναι αλληλένδετα, πάνε χέρι-χέρι και χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πώς να εξηγιάνεις ένα προπολογισμό. Και αν δεν έχεις εξηγίαση του προπολογισμού είναι δύσκολο να τονώσεις την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχουμε πλήρη επίγνωση εμείς αυτών των προκλήσεων του στρατηγικού αυτού τριγώνου. Και πολιτικά είναι πολύ σημαντικότερα αυτά από την καταπολέμηση της κρίσης αυτής καθ' Κάποτε είπα στο κοινοβούλιο μας ότι πολιτικά μπορεί πιο εύκολα να συμφωνήσει κανείς να δαπανίσει μερικά δισεκατομμύρια παραπάνω αλλά είναι δύσκολο να συμφωνήσει πολιτικά για το πώ θα συμμαζέψει τον προϋπολογισμό σου. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, τα αναγνωρίσουμε όλα αυτά. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και η Ευρώπη ως ε, τόπος οικονομικής παραγωγή, οικονομική δραστηριότητα. Γιατί έχουμε την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη σάντουιτς. Θα την ε, συνθλίψουν οι Ηνωμένε Πολιτείε η Βραζιλία από τη μια και η Ασία από την άλλη. Η Ευρώπη είναι στη μέση. Ε, για την Αυστρία, για τη δική μας οικονομική πολιτική, αυτό το στρατηγικό τρίγωνο είναι τμήμα της εθνικής πολιτικής. Έχουμε κάποιους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ήδη προεξοφλήσει. Ήδη από το έτος 2007 αποφασίσαμε αλλαγή ε, του δικαίου προϋπολογισμού και χρειάστηκε και αναθεώρηση του συντάγματος. Από το ε, νέα άρχισε η πρώτη εφαρμογή, η πρώτη φάση και η δεύτερη ακολουθήσει το 2013. Για τα επόμενα λοιπόν τέσσερα έτη κάθε φορά ορίζουμε ένα πλαίσιο με οροφές για όλες τις δαπάνες ε, και είναι μια τροχοπέδια, ένα φρένο για τις δαπάνες βλέπε, και φρένο για το χρέος τελικά. Και κάθε χρόνο ε, προστίθεται ένα νέο έτος για να γίνει τετραετία. Φέτος είμαστε στο 2014, από του χρόνου θα κάνουμε μέχρι το 2015. Λοιπόν, αυτή η οροφή των δαπανών παντού ε, συνδέεται με μεγαλύτερη ευελιξία. Εάν υπάρχει κάποια δυνατότητα ε, σε ορισμένες δαπάνες μεταφέρονται πιστώσεις σε άλλες που δυσκολεύονται περισσότερο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία πάρα πολύ χρήσιμη. Το 2013 θα έχουμε μια τελείως καινούρια δομή. Ε, ε, η λογιστική μας ε, θα περάσει σε πιο εμπορική λογική αν θέλετε από την αρκετά σφιχτή αμυγός λογιστική και θα προϋπολογίζεται και το θέμα του φίλου, το gender budgeting. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες αλλά χρειάζονται και προγράμματα εκπαίδευσης αλλά ε, το διαχωρίζουμε το ένα σκέλος της κατάρτισης του προπολογισμού είναι στο Υπουργείο Οικονομικών και ε, ένα άλλο σκέλος ελέγχου είναι στην Καγκελαρία, είναι σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Ε, το έλλειμμά μας ήταν 4,1 πέρσι, 3,2 φέτος και για το χρόνο φιλοδοξούμε 2,9%. Νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά για την πρόκληση αυτή. Φέτος τον Απρίλιο η κυβέρνηση θα υποβάλει το πλαίσιο το δημοσιονομικό για την επόμενη τετραετία. Θα το συζητήσουμε και στο Κοινοβούλιο και για την Αυστρία θα τα διαβιβάσουμε και αυτό το σύμφωνο σταθερότητα στην Ευρώπη. Ξέρετε, έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητα στην Αυστρία μεταξύ του κράτου, των ομόσπονδων κρατηδίων και των δήμων και κοινοτήτων. Όλα τα κράτη πρέπει να κάνουν προπολογισμού ε, ε, οικονομία, ε, εξοικονομήσουν χρήματα και δαπάνε, αλλά θα ήταν χήμερα να πιστέψει κανεί ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να διευρυνθεί, να μεγεθυνθεί. Είναι μοναδική σήμερα η ευκαιρία. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο-τρει χώρε που διαφωνούν, ε, αλλά θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος χρηματοοικονομικές συναλλαγές, γιατί ε, έχει αποσυνδεθεί πλήρως αυτός ο κλάδος της οικονομίας, ο χρηματοπιστωτικός, ε, από την πραγματική οικονομία. Το είπαμε και προηγουμένως. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Ε, έχουμε και θέματα μισθών, θέματα συντάξεων που είναι επίμαχα αλλά θα πρέπει και οι κοινωνικοί εταίροι να στραφούν στην παραγωγικότητα. Και επίσης το ε, όριο ηλικίας συνταξιοδότηση θα πρέπει να προσανατολίζεται στην ηλικία του πληθυσμού. Τελειώνω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι, επαρκές, δεν είναι αρκετό να έχουμε μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο τέτοιου είδους ε, συνεδριάσεις. Νομίζω χρειάζεται σε πιο τακτά ε, χρονικά διαστήματα να κάνουμε κοινέ συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ακολουθούν οι συγητές μας για τη δέσμη ε, διακυβέρνησης που ονομάζεται Six Pack. Πολύ αρενοπή αυτή η έκφραση. Ο κύριος Φέο πρώτος. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε αυτή τη συνεδρίαση. Κατά τη διάρκεια έξι χρόνων ε, διατέλεσα εθνικό βουλευτής και διαπιστώνω σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση μια τροποποίηση σε σχέση με την ε, ε, τον τρόπο αντιμετώπισης των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, των Εθνικών Ζητημάτων, συζήτησης των Ευρωπαϊκών Θεμάτων και κατανοούν και τη σημασία των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Μέσα αυτό το πακέτο των ε, νομοθετικών προτάσεων περιλαμβάνονται κάποιες καινοτομίες. Αυτές έχουν ως βάση τα προηγούμενα την προέλευση της κρίσης και τη δυσκολία που αντιμετώπισαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, και γι' αυτό και θεωρώ ότι, ότι για να γίνει πιο αξιόπιστο το σύμφωνο αναπτύξης και σταθερότητας ήταν απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια πιο έντονη μορφή στο κριτήριο του χρέους και θεωρώ πως είναι σκόπιμο επίσης να ε, υπάρξει μια συγκεκριμένη διαδικασία όσον αφορά την μακροοικονομική ισορροπία, να θεσπιστούν νέες διαδικασίες στους τομείς του προπολογισμού και επίσης ε, Θεωρώ πως είναι απαραίτητο να υπάρξει και ένα σύστημα κινήτρων που να συνοδεύει το σύστημα των κυρώσεων. Το Κοινοβούλιο συζήτησε, ε, μάλιστα υπήρξαν καινοτόμες ιδέες με τους, ε, συζήτηση με τους συζητητές και το Κοινοβούλιο ε, δεν ε, θα πρέπει να δεχτεί απλά τα όσα παρουσιάστηκαν. Θα πρέπει να γίνουν συζητήσει επίκαιρε. Θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να συνοδεύσουμε τα όσα λέγονται εκτό του Ευρωκοινοβουλίου και όταν θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η εργασία, το Κοινοβούλιο θα έχει ω θεσμό το δικό του λόγο ανεξάρτητο λόγο σε σχέση με αυτά τα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο παίζει κεντρικό ρόλο μέσα στο πακέτο αυτό Και επειδή εδώ είμαστε σε ένα θεσμικό πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ένας ε, πολύ καλός στόχος. Δεν ε, θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο με τα, για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να μιλήσουμε και για τους στόχους. Και γι' αυτό και το σύμφωνο σταθερότητας θα πρέπει να είναι όλα και περισσότερο σύμφωνο ανάπτυξης. Ε, ε στα και ποιοι θα είναι οι στόχοι σε διάφορα κράτη. Η απάντηση στην κρίση με πακέτα λιτότητες δεν αρκεί. Θα είναι απαραίτητο να δούμε ποιε είναι οι προοπτικές που υπάρχουν στις οικονομίες, για τις οικονομίες μας. Τι εμείς ε, υποστηρίζουμε. Γιατί, ναι, πρέπει να μπει τάξη στην δημόσια οικονομία, να λιμιωθεί το έλλειμμα, αλλά για αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια προοπτική για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας που θα δέχεται τις διαφορετικές πραγματικότητες, τις διαφορετικές ανάγκες κάθε οικονομίας. Μένες οικονομίες χρειάζονται περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές, άλλες ε, συγκεκριμένες ε, ε, ενέργειες σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά και γι' αυτό ακριβώς και χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η εφαρμογή της κοινοτικής μεθόδου. Και επίσης, για τον ίδιο λόγο, σε αυτήν την ε, φάση οι λύσεις είναι δύσκολες και πρέπει να ε, μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και ολοκληρώνω αναφερόμενο στο, λόγο, στο, στο ρόλο συγγνώμη, των Ευρωβουλευτών και των βουλευτών γενικότερα. Θα πρέπει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λειτουργήσει εντατικά. Δεν είναι λογικό έγγραφα όπως το τα σταθερότητα και ανάπτυξη που υποβάλλονται στις Βρυξέλλες να μην συζητώνται στα εθνικά κοινοβούλια. Όχι μόνο πρέπει να συζητηθούν, αλλά ίσως και ακόμα, ακόμα και να ψηφιστούν στα εθνικά κοινοβούλια. Όχι μόνο θα πρέπει να είναι έγγραφα τα οποία παραδίδουν στις Βρυξέλλες οι κυβερνήσεις χωρίς να προβαίνουν στην απαραίτητη προηγούμενη εσωτερική συζήτηση. Νομίζω πως και αυτό είναι τμήμα καλύτερου συντονισμού. Θα πρέπει να δούμε κοινά σημεία και άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όλο ένα και περισσότερο μετατρέπεται σε ένα κοινοβούλιο όπου ε, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ε, ρόλο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η Ελίζα Φερέιρα τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ θα ξεκινήσω εκεί ακριβώς που σταμάτησε ο συνάδελφος Διέγκο Φέιο. Εγώ πιστεύω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα μέσο ε, πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσει να προωθήσει το συντονισμό ανάμεσα στα προγράμματα των διαφόρων χωρών και έτσι ώστε εντός κάθε χώρας να μπορέσει να υπάρξει συνέπεια, συνοχή ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στους εθνικούς μας στόχους. Δεν μπορούμε να μετατραπούμε σε ένα μέσο επιβολής οδηγιών, ευρωπαϊκών οδηγιών ούτε μπορεί να αποτελέσει μέσο που θα θα, θα πάρει την στρατηγική και την ευθύνη για τη στρατηγική από κάθε χώρα. Αν χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο αυτό το μέσο θα είναι αρνητικό στην εφαρμογή του. Τώρα όσον αφορά τη νομοθετικά κείμενα επί των οποίων ε, από κοινού εργαζόμαστε, θα αυτό που αποτελεί μια ευκαιρία ιστορική σημασία θα έλεγα για να εισάγουμε μεγαλύτερη, περισσότερο ορθολογισμό, ρεαλισμό και αποτελεσματικότητα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το να έχουμε από κοινού μια ανάλυση του, του ελλείμματος, του χρέους και των ε, μακροοικονομικών αρισορροπιών είναι κάτι θετικό. Όμως, ε, έχουμε επίσης εδώ, διατρέχουμε τον κίνδυνο να μετατρέψουμε το μέσο αυτό σε ένα πακέτο και το κυρώσεων. Και αυτό δεν θέλουμε να συμβεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μετατρέψουμε αυτά τα νομοθετικά κείμενα σε μια τυφλή ε, τιμωρία για τη χρέος, το έλλειμμα και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Και άρα... Το Κοινοβούλιο θα προσπαθεί να βελτιώσει και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε, να βελτιώσουμε λοιπόν τις προτάσεις που επέβαλε η Κομισιόν. Υπάρχουν κάποια άξονες επί των οποίων αρχίζει να προκύπτει κάποια συνένεση. Ε, μία, ένας από αυτούς είναι ότι μέσα σε αυτή τη ε, νομοθετική διαδικασία στις διάφορες φάσεις εφαρμογής είναι σημαντική η συμμετοχή των εκπροσώπων των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ορισμένες φάσεις των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ είμαι η συγχύτρια για το καινούριο νέο στοιχείο που είναι το στοιχείο των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Είναι ένα κείμενο στην απόφαση και πιστεύω ότι για να είναι χρήσιμο θα πρέπει να συνδυαστεί με κάποιο πολύ στενό τρόπο με τα νέα στοιχεία τα οποία έρχονται τώρα στη συζήτησή μας μέσω του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας, του Συμφώνου για το Ευρώ. Δηλαδή, όταν αναλύουμε την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων χωρών, χρειάζεται να καταφέρουμε να συνδυάσουμε αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή με μια διακυβερνητική βάση με το νέο στοιχείο στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και το αποκαλούμε μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την ερμηνεία και την ερμηνεία που δίνεται στο επίτευξη της μείωσης του ελλείμματος ή του χρέους, να κατανοήσουμε ποια είναι η ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας, να δούμε πώς κινείται η πραγματική οικονομία, η ανάπτυξη και η απασχόληση, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την βιωσιμότητα, την μακροπρόθεσμη αυτών των ε, ευαίσθητων ισορροπιών, που είναι απόλυτα ονομαστικού χαρακτήρα. Έπειτα, Άλλο σημείο που υπάρχει κάποια πρώτη συνένεση είναι αυτό το πλαίσιο των μακροοικονομικών διαφορών ε, το θέμα των κυρώσεων και των προστήμων. Μια χώρα δεν μπορεί να τιμωρηθεί επειδή δεν καταφέρει να φτάσει σε περίπλοκους ε, στόχους. Ε. Θα μπορεί μόνο να τιμωρηθεί αν δεν έχει καταβάλει την απαραίτητη προσπάθεια που χρειαζόταν για να επιτύχει τους στόχους αν έχει στάση αρνητική δεν είναι συνεργάσιμη γιατί ο, οι στόχοι μακροοικονομικοί είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και δεν μπορούν να ερμηνεύονται με απόλυτο και τυφλό τρόπο. Οι ευθύνε που βαραίνουν κάθε κράτος θα πρέπει να εξεταστούν με συμμετρικό τρόπο Δηλαδή, οι χώρες που έχουν ε, λίμα και οι χώρες που έχουν πλεόνασμα θα πρέπει να συζητήσουν τις στρατηγικές τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δείκτες είναι αυτόματοι. Θα πρέπει να προτείνουν μια πιο λεπτομερή ανάλυση της διασύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες κρατικές οικονομίες. Συνοψίζω, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιο είναι το περιθώριο ελιγμού κάθε χώρας, το πραγματικό και ποιο είναι το περιθώριο ελιγμού που έχουμε γενικότερα. Γιατί οι ευρωπαϊκέ οικονομίε είναι τόσο συνδεδεμένε μεταξύ του που ορισμένε ενέργειε σε μήνα κράτου μπορεί να έχουν επιπτώσει στην οικονομία άλλου κράτου. Ε, νομίζω λοιπόν πως είναι τεράστιο το δυναμικό για ευρωπαϊκή πρόοδο. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το χώρο το, που μας ανοίγεται μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ πέρα παρόντες, ταξιδεύσατε ε, εδώ για να συζητήσουμε όλοι μαζί. Υπάρχουν δύο λόγοι για το ότι πρέπει να δουλέψουμε από, από κοινού. Υπάρχει η νομική πτυχή και ο άλλος λόγος είναι η, η κρίση. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας όλα είχαν ενισχυθεί. Έχουν μεγαλύτερο λόγο τα εθνικά κοινοβούλια και επίσης όλα είχαν διαβρεθεί. Αλλά τα κοινοβούλια θέλουν απλώς να κάνουν το έργο τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να έχει τις δικές του ευθύνες, ευθύνες στις οποίες, α, ε, οποίες του δόθηκαν από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όταν διαβάζετε τα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όλα θα αποφασιστούν τέλη Μαρτίου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Φανερουμπόη υπογράμμισε ότι είχε γίνει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσιονομικών και το Κοινοβούλιο βοήθησε ε, κάπως τα, τις χώρες μέλη για να πάρουν αποφάσεις. Έχουμε λοιπόν μια κοινή ευθύνη και η οποία είναι σοβαρή. Η δική μας ευθύνη είναι ότι όσο δυνατόν πιο γρήγορα, σε μήνες, χρόνια, να κοιτάξουμε να δώσουμε μια ελπίδα, ελπίδα στους Ευρωπαίους. Αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρε μέλη υπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και εμεί θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, που δημιουργούν μια αλληλεξάρτηση. Έχουμε μια διάγνωση σε ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τι έχει συμβεί. Για την Ευρωζώνη λέω τώρα. Έχουμε χώρε μέλη ε, οι οποίες δεν σεβάστηκαν τις δεσμεύσει τους ούτε για τα θέματα πειθαρχία, δημοσιονομική πειθαρχία, ούτε σε θέματα ανταγωνιστικότητα. Υπενθυμίζω, ακόμα και αν είχαμε την ανοιχτή ε, μέθοδο συντονισμού, ε, θελήσαμε σε, πιο, σε υψηλό επίπεδο να κάνουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι ε, το περισσότερο δυνατό ανταγωνιστική. Επίσης, να πω ότι είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν αρκεί κάθε χώρα να κάνει αυτό που υποτίθεται ή που θεωρεί ότι κάνει το θέμα που έχουμε μπροστά είναι το εξή. Πώς θα διασφαλίσουμε ούτω ώστε να έχουμε ένας ε, αμοιβαίος έλεγχος ε, με την καλή έννοια, όχι αστυνομικό έλεγχο, ούτω ώστε να προβλέψουμε, να προλάβουμε μάλλον, τι, αν υπάρχει κάτι το οποίο πάει να ε, εκτροχιαστεί. Δι, αν δεν το πετύχουμε αυτό, χάσαμε. Θα πρέπει να δούμε επίση πώ μπορούμε αμοιβαία να ασκήσουμε μια πίεση. Και εδώ θα πρέπει να δούμε δηλαδή κάτι το οποίο είναι σημαντικό, αλλά όχι ότι έρχεται να υποκαταστήσει τα, τα, τις εθνικές ευθύνες. Έχουμε το σύνολο του πακέτου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ειλικρινή διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν κάνει μια έκθεση η Επιτροπή για την κατάσταση σε μια χώρα, για τα δημοσιονομικά της, τα μακροοικονομικά της, εμείς αυτό που θέλουμε είναι όχι εξουσία, αλλά ένα διάλογο ο οποίος μπορεί να λάβει υπόψη τις συνέπειες σε σχέση με τις αποφάσεις που έχουν ελευθεί στην ΑΒ χώρα. Σε θέματα που είναι μισολογικά, ε, ε, συντάξεις, απασχόληση, χρειαζόμαστε ένα διάλογο ο οποίος είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, πέρα από τα σύνορα, πέρα από γλωσσικά φράγματα. Αυτό είναι η πρότασή μας. Να το δείτε λοιπόν, να τη δείτε την πρόταση. Όχι ότι μια ε, επιθυμία να αποκτήσει εξουσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον κύριο Παπανδρέο είχαμε πέρσι μια συνάντηση. Και είναι σημαντικό που ένας, ε, κάποιος ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μια χώρα, υπεύθυνο. Χρειαζόμαστε αυτό το διάλογο. Ήρθε εδώ να μιλήσει μαζί μας. Και θα κλείσω. Τώρα, αυτή είναι η πρόταση που κάναμε. Δεν έχουμε ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή μας, δεν είχαμε απόφαση του Κοινοβουλίου, αλλά όπως αναφέρθηκε να πω ότι εμεί και κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί την, ε, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί τη θέση που έχει το ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουμε μόνο τι σχέσει ανάμεσα σε ευρωπαϊκέ χώρε. Έχουμε ένα ε, νόμισμα το οποίο είναι δυνατό σε παγκόσμιο επίπεδο και όπω είπε και ο κύριο Φανορομπόη, ε, το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε και όταν μακροπρόθεσμα εξηγιάνουμε τα οικονομικά μας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να μπούμε στον κόσμο με ε, ε, αισιόδοξα και αποφασιστικά. Ας δούμε τι ακριβώς γίνεται στις άμα δει κανεί πώ έχουν κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, το, Ευρωπαϊκ... το ευρώ δεν δε χρειάζεται να κοκκινίζει. Ευχαριστώ. Κυρία Φόρτ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τα, τους εθνικούς βουλευτές να μας περιγράφουν τι ε, κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση τα κράτη της. Για μένα, στη δέσμη ε, της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε υγιείς οικονομίες στα κράτη-μέλη. Αυτό έχουμε ως στόχος. Και να καταλάβουμε ότι η υγεία ενός κράτους επηρεάζει την υγεία άλλων κρατών. Ε, και οι μοίρες μας είναι συνδεδεμένες, σε κάποιους τομείς περισσότερο, σε κάποιους άλλους λιγότερο. Και έχουμε όλοι συμφέρον να είναι υγιής οικονομία. Ε, προηγουμένως η Σόφη Νετβέλτ μίλησε για 27 χώρες που θα πρέπει να καταλήξουν να φάνε το ίδιο σάντουιτ το μεσημέρι. Μα μπορεί κάποιο να έχει γίνει διατροφή ω χώρα χωρί να είναι υποχρεωμένο να τρώει την ίδια τροφή με όλου του υπολείπου. Δηλαδή, αυτό το θέμα που ονομάζεται ownership, δηλαδή κάθε χώρα ε, έχει το δικό της τρόπο να αντιμετωπίζει την κατάσταση και να βρίσκει εκείνη ποια είναι η υγιεινή διατροφή που της ταιριάζει. Και όχι μόνο βράχει πρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Αυτό ε, θα το βρείτε και στην διέκθεσή μου για το πλαίσιο, για τη διαφάνεια, για τα χρήματα των φορολογουμένων ε, και διαφάνεια και προς τα άλλα κράτη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική σας το σχεδιασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να βλέπουμε πόσο ρευστό έχει η τράπεζα ας πούμε και να καταλαβαίνουν και ε, πώς φτιάχνουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όλοι. Καταλαβαίνω επίση ότι ο καθένα θα πρέπει να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Γι' αυτό μιλάμε για εθνικού, αριθμητικού κανόνε που εφαρμόζει η κάθε χώρα. Ερχόμαι τώρα στη δημοφιλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι πολύ συχνά όταν κάποιο σου παίρνει τι σοκολάτε και τι καραμέλε, ε, είναι πάρα πολύ αντιπαθής. Ε, γι' αυτό και τώρα που έχουμε λιτότητα, το Συμβούλιο έχει το ρόλο του, δεν είναι μόνο τα θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, μας ε, παίρνουν τα γλυκά. Είναι και οι χώρες. Α, και επίσης ποιος έχει προσκυκληθεί ε, Προσκληθεί, συγγνώμη, στο γεύμα αυτό είναι 17, είναι 27, είναι 17 συν όσοι θέλουν να μπουν στο ευρώ. αυτό συμπεριλαμβάνει ή αποκλείει το Ενωμένο Βασίλειο. Πώς γίνεται η πρόσκληση σε αυτό το γεύμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνδεσης διαφόρων οικονομιών. Βεβαίως, εκείνοι που συμμετέχουν στο ευρώ έχουν απεμπολίσει κάποια φάρμακα που θα μπορούσαν ε, να χρησιμοποιήσουν για να επανέλθουν στην υγεία, γιατί έχουν κοινό νόμισμα. Ο συνάδελφος από την Πολωνία ήταν πολύ σαφής αυτά που είπε Αναγνωρίζω επίση αυτά που λέτε για τα θέματα των συντάξεων και τι συνταξιδοτικές μεταρρυθμίσει. Η αλλαγή των κανόνων για χώρε που προσπαθούν να πάρουν το φάρμακό του για να λύσουν το πρόβλημα και να επανέλθουν. Ε, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό να είναι μόνο βραχυπρόθεσμη μια στρατηγική. Και συνεχίζοντας αυτή την αναλογία, ποιο είναι το αίτιο της ασθένειας. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε ο Βέλγος συνάδελφος για τη Βασιλεία και τις Τράπεζε. δεν είναι μόνο ε, το κρατικό χρέος, το δημόσιο χρέος, αλλά πολλές φορές και το ιδιωτικό ε, χρέος, ε, υπερβολική δανειοδότηση των τραπεζών σε αφαιρέγγιους δανειολήπτες που οδήγησε αυτή τη φούσκα. Η Northern Rock, θυμάστε, μια μεγάλη εμπορική τράπεζα που είχε μαζική ανισορροπία ε, στη ρευστότητα. Δεν ήταν επενδυτική τράπεζα, ήταν ε, μια τράπεζα που είχε πρόβλημα στη ρευστότητα, στις κεφαλαϊκές απαιτήσει και που υπερδανειοδότησε ε, δανειολήπτες που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν τα δανειά τους στο G20 η Γαλλία θα πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, πρωταγωνιστικό. Ας μην θεωρήσουμε ότι τα τραπεζικά προβλήματα δεν υπήρξαν στην Ιρλανδία, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία. Ήταν το θέμα των πιστώσεων, ήταν το θέμα της ρευστότητα και γενικότερο θέμα των τραπεζών. Πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωρούμε τώρα στη συζήτηση. Ε, θέλετε, Γενική, έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να σας διαβάσω τα ονόματα, έτσι για να γνωρίζετε. ζοζέτη από την Ιταλία, Βοσκάνη από τη Ρουμανία, από τη Γαλλία, Γκομπέρ, δεν ξέρω αν κύριος ή κυρία, ο κύριος Ανδριοκάτης από τη Λιθουανία, από την Ιταλία και πάλι έχω τον κύριο Καραβάλια και από τη Λετωνία Κρίξ νομίζω και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα ο Σουζέ Μανουέλ Καρσία Μαργάγιο. Ο κύριος Τζορτζέτσι παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς στο Ιταλικό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε να δεχτούμε τις υποδείξεις όσο γινόταν πιο γρήγορα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και πιστεύουμε ότι μέσα σε δύο-τρεις εβδομάδες θα το εντάξουμε στην εθνική μας νομοθεσία τα όσα μας υπέδειξε το ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιολογούμε θετικά και αυτή την κατεύθυνση που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της στρατηγικής 2020 και να τις μετρήσουμε με ποσοτικούς όρους. Ε, ωστόσο είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η εξαιρετικά φιλόδοξη στόχοι κατά κάποιο τρόπο δεν θα πω ότι είναι αλλά είναι ένα trade-off σε σχέση με τους στόχους ε, μείωσης του ελλείμματος και του χρέους και νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν αυτές οι δύο θεμητές ε, προσδοκίες. Εμείς ως Επιτροπή Προπολογισμού εξάλλου είμαστε συνηθισμένοι τα τελευταία χρόνια να συνοδεύουμε την κυβέρνηση στην πειθαρχία, τη δημοσιονομική και όχι σε δραστήριες πολιτικές οικονομικής ανάκαμψης και γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να τονίσουμε δύο πτυχές ότι εν μέσω όλων αυτών των δυσκολιών υπάρχουν δύο θετικές πτυχές. Πρώτον, εμβάθυνση ε, που είναι αυτά τα σχέδια, τα εθνικά σχέδια μεταρρύθμισης που θα πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο πριν από την υποβολή του προγράμματος στην Ευρώπη μας, μας υποχρεώνουν να εξετάσουμε τις μεγάλες πολιτικές, ε, τις οικονομικές πολιτικές όσον αφορά την ανάπτυξη και την ε, εξέλιξη. πρώτη φάση, όπως ήδη τόνισε και ο Γάλλος συνάδελφος, το περασμένο χρόνο η συζήτηση ήταν ε, πολύ βιαστική ενώ όσον αφορά την οριστική οθέτηση που προβλέπεται για τον Απρίλιο, εμείς ε, ερχόμαστε σε επαφή με όλες τις οικονομικές κατηγορίες, με όλους τους μεγάλους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας για να συζητήσουμε ακριβώς το εθνικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης. Αυτό δεν είχε γίνει πριν και αυτό σίγουρα γίνεται χάρη στα κέντρα και τις υποδείξεις της ευρωπαϊκές. Δεύτερο θετικό στοιχείο που ήθελα εγώ να αναφέρω και επαναλαμβάνω ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες δεν ε, παραγνωρίζουμε αλλά η θετική, θετικό στοιχείο είναι αυτή η δύσκολη ανταπαράθεση που ωστόσο εντάσσει τα εθνικά μας κοινοβούλια σε μια συζήτηση από τα οποία παλιότερα αποκλειόταν τελείως. Η συζήτηση γινόταν ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εμείς έπρεπε δηλαδή απλώς να μετατρέψουμε σε εθνική νομοθεσία κάτι διαπραγματεύσεις από τις οποίες τελείως ε, αποσιάζαμε. Τώρα είμαστε μέρος τη συζήτησης, εντάξει δεν καθορίζουμε εμείς τη γραμμή αλλά κατά κάποιο τρόπο συμμετέχουμε. Και πιστεύω πως ακριβώς αυτή η φάση συζήτησης θα μπορούσε να γίνει κάπως νωρίτερα ώστε να εντοπιστούν οι καλύτερες πρακτικές και να προσπαθήσουμε να τις ε, οικειοποιηθούμε. Εντάξει, είμαστε ένα σωρό χώρε, 27 χώρε, η καθεμιά με την ιδιαιτερότητά τη. Αλλά είναι στιγμέ δύσκολε που σίγουρα με τον καιρό θα φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Και έπειτα στη συνέχεια σίγουρα θα βελτιωθούν τα πράγματα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Από τη Ρουμανία τώρα, ο κύριος Φαλσκάνη. Ευχαριστώ πολύ στα αγγλικά. Καταρχάς θα ήθελα να σας εκφράσω την άποψη της ε, ρουμανικής γερουσίας. Εμείς θέλουμε να ε, διατηρηθεί και να διευρυνθεί η συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάρα πολύ σημαντικό για να φτάνουμε από κοινού στους στόχους της εθνικής του 2020 και την οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα όμως με κάθε σεβασμό για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, είναι τρία τα ζητήματα. Διαδικαστικά, τεχνικά, δεν έχουμε συζητήσει τίποτα τεχνικό ακόμα και τους τομείς που όλα αυτά εφαρμόζονται. Πρώτον, τα διαδικαστικά. Γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέτουμε σε διαφορετική βάση ε, τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τις χώρες μέλη. Άλλη σχέση έχουμε εμείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε τα μακροοικονομικά μας επίπεδα, τα εθνικά και την εσωτερική στρατηγική και τις παραδοχές που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε επικάλυψη. Αυτό το κάνουμε ήδη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το δεύτερο, τεχνικό ζήτημα. Ποιοι είναι οι μακροοικονομικοί δείκτε που λαμβάνουμε υπόψη. Γίνεται στο G20 τώρα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το συνδυασμό των ε, στοιχείων ε, του δημοσίου χρέους και του εξωτερικού χρέους με το εσωτερικό ε, και πώς είναι το επίπεδο καταθέσεων και αποταμιεύσεων του πληθυσμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε τι κριτήρια χρησιμοποιούμε στο μέλλον για να δημιουργούμε μοντέλα τέτοια για τα κράτη μας. Άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι σημασία έχουν οι διάφοροι δείκτες στη χώρα μου, ο δείκτης ενεργείας δεν έχει καμία σημασία, διότι ο μισός πληθυσμός είναι τελείως εκτός αγοράς εργασίας. 20% είναι στη Γεωργία περίπου, 20% είναι διασκορπισμένοι ανά την Ευρώπη κτλ. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν και πού συνεργαζόμαστε. Ας πούμε τα συστήματα υγείας το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τα ταμεία. Όλα αυτά δεν είναι σήμερα τμήμα της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής και θα πρέπει να γνωρίζουμε σε τι βάθος έχει γίνει η ανάλυση των στόχων αυτών. Και ένα τελευταίο όπου θα ήθελα να θέσω υπόψη σας είναι η προβλεψιμότητα. Αν αλλάξει κάτι κατά τη διάρκεια του έτους, δεν μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε τα ίδια συμπεράσματα των συζητήσεων του Απριλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν χώρες σαν μου με μια οικονομία πάρα πολύ δυναμική. Ευχαριστώ. Από τη Γαλλία τώρα, ο κύριος ή η κυρία Γκομπέρ, δεν ξέρω. Non, Okay, thank you. <laughs> Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου εντάσσεται σαν σα απαντήσει στην ομιλία του κύριου Φαναντεμπόη. Εγώ συμμερίζομαι αυτά που είπε, που είναι διαφορετικά αυτά που διαβάζει κανείς, δηλαδή τους στόχους για θέματα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά τα μέτρα που μπορεί να έχει κανείς στη διαθέση του, αυτά είναι κάτι που μπορούν να συζητηθούν. Σύντομα όμως να αναφέρουμε κάποια πράγματα. Όταν μιλάμε για μέσα μιλάμε για τους προϋπολογισμούς και αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με άλλες χώρες που είναι πολύ αδύνατες φέρει Πολύ λίγοι δέχονται ε, πολύ λίγοι θέλουν να συζητάνε το θέμα της μείωσης των φόρων και η Αγκαλία είναι το παράδειγμα που το έχει κάνει και δεν οδήγησε σε κάτι αρνητικό. Φυσικά το θέμα της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων είναι σημαντικό. Επίσης έχουμε να κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίε. Πώς θα γίνει, μήπως πρέπει να έχουμε ε, ή όχι ιδιωτικοποιήσεις. Ε, κατάρτιση, που μπορεί να, αν είναι ιδιωτική ή όχι, εκπαίδευση και αυτό μπορεί να επιβαρύνει την, ε, τα, τα οικονομικά των οικογενειών. Ε, δεν γίνεται αναφορά λοιπόν σε όλα αυτά. Και όπως ανέφερε ε, η Σύτρια Βρετανή, ε, είναι θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Έχουμε φέρει πίν πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν, είναι καταχρωμένες και τους δίνονται, τους, τους προτρέπουν να έχουν κουράγιο κτλ. αλλά δεν έχουν τα μέσα να ανταπεξέλθουν. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Διατροφή, εκπαίδευση, όλα αυτά. Το θέμα είναι το θερμόμετρο που έχουμε για να κάνουμε μια αξιολόγηση είναι σωστό σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα. Γίνεται δηλαδή σωστή αξιολόγηση. Να το δούμε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Χωσέ, θες να μιλήσεις τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος. Θα ήθελα να θυμίσω ε, τα εξής αρχικά. Ο κύριος Τρισέ, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ε, ε, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση. Τις θεωρεί πολύ αδύναμες και πολύ ασθενείς και θεωρεί ότι θα τις είχε αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο το Συμβούλιο και αναλογεί τώρα στα Εθνικά Κοινοβούλια μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανορθώσουν. Τι συμβαίνει τώρα. Όλα τα θεμέλια στα οποία βασίζεται ή βασιζόταν εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν ή ο ναι, κατέρευσαν ή καταραίων. Τρία ήταν τα θεμέλια αυτά. Όχι διάσωση, no bailout, no default, no exit. Τώρα έχουμε bailout με τη διάσωση, τον προσωρινό που θα γίνει οριστικός μηχανισμός. Το no default επίσης έχει αλλάξει με το μόνιμο μηχανισμό που ε, θα ε, συμμετάσχει και ο ιδιωτικό τομέας και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε νέο έδαφος, άγνωστο έδαφος, τέρα incognita. Και έχουμε μεταβλητές που δεν γνωρίζουμε. Αυξάνεται η δημοσιονομική πειθαρχία και η ανταγωνιστικότητα, καλό αυτό, και ένα μηχανισμό διάσωσης έχουμε πλέον μόνιμο και διαρκή με ιδιωτική συμμετοχή, που και αυτό μπορεί να είναι συζητήσιμο, αλλά υπάρχει. Στο προσωρινό μηχανισμό διαπιστώσαμε ότι απέτυχε. Το είδε και το Κοινοβούλιο. Στις 11 Μαρτίου αποφασίστηκε να μειωθεί το επιτόκιο για την Ελλάδα και ζητάνε από την Ιρλανδία να κάνουν κάτι με τους φόρους τους για να μειώσουν και σε αυτούς το επιτόκιο. Με τέτοια επιτόκια πού να αναπτυχθεί κανείς και χωρίς περιθώριο για την ανάπτυξη δεν μπορεί να ε, μειωθεί το χρέος. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ενδιάμεσος μηχανισμός που είναι τα περίφημα ευρωομόλογα δεν είναι όμως αυτό ο μηχανισμός για χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχία και μπορούμε να συζητήσουμε και το ποσοστό του χρέους που θα μπορεί να ληφθεί χωρίς να διακυβευτεί η σταθερότητα της Ευρωζώνης. Επίσης, είμαστε διατεθειμένοι να δούμε και τη δυνατότητα της πρόσβασης του συνολικού ταμείου. Οι ευρωπαϊκές χώρες να συνδέουν τη συμπεριφορά τους με την προσφυγή. Οι χώρες που είναι λιγότερο ενάρετες στην αρχή και βεβαίως να πληρώνουν κάποιο επιτόκιο επιπλέον. Αυτή την πρόταση την έκανε και η ίδια η πρόεδρος και σε μια δεύτερη φάση, αν συνεχίζουν στη μη συμμόρφωση, ε, να μην ε, έχουν τη δυνατότητα ψήφισης ποσόστησης και τέλος να υπάρχει δυνατότητα ε, πλήρους απόκλησης τους από το μηχανισμό αυτό. Και έτσι λοιπόν θέλω να τονίσω το εξή. Μεταξύ της δημοσιονομική πειθαρχίας και του μονίμου μηχανισμού λείπει μια ενδιάμεση γέφυρα, ένα συνδετικός κρίκος. Για να μην προσφεύγουμε συνέχεια στο μηχανισμό αυτό που δεν θα λειτουργήσει. Και επίσης να τονίσω ότι τα ευρωομόλογα δεν είναι ένας μηχανισμός ε, εγκατάλειψης, χαλάρωσης της πειθαρχία, αλλά ένας αυτόματος μηχανισμός ακριβώς ε, να εγγυηθούμε αυτή την πειθαρχία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Λιθουανία πάμε τώρα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι συζητήσεις μας έχουν να κάνουν με το διάλογο ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτού του διαλόγου θα πρέπει να συμμεροζόμαστε ε, κάποια συγκεκριμένα θέματα και βλέπω όμως τώρα συζητάμε για τα πάντα και γενικά. Υπάρχουν ε, πολύ συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε στη Λιθουανία στα πλαίσια της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Υπόθεσεις και με τις ε, Επιτροπές για τα ε, Οικονομικά έχουμε κάνει κοινέ ε, συνεδριάσεις και διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε χρόνο κατάλληλο για να οργανώσουμε αυτό το διάλογο. Τα θέματα είναι, τα έγγραφα είναι πολλαπλά. Μας είπανε πριν από το Φλεβάρι υπάρχει το πρόγραμμα το ε, για τους ε, εθνικούς δείκτες, άλλα προγράμματα και ανα... έπρεπε να έχουμε αναλύσεις εγγράφων πριν από το Φεβρουάριο. Είχαμε τόσα πολλά έγγραφα και δεν ήταν εύκολο να προχωρήσουμε. Πριν από το Μάρτι πιστεύουμε ότι θα έχουμε, μια θα έχουμε κατευθύνες γραμμές για την ε, δημοσιονομική πολιτική και μετά πριν από τον Απρίλη θα έχουμε το γενικό πλαίσιο που αφορά το πρόγραμμα σύγκλησης. Το Μάιο θα έχουμε το νομοσχέδιο ε, εκ μέρους της Ευρω... Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν τόσα και τόσα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε με τις αρμόδιες επιτροπές, τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να έχουμε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα. Ίσως αυτό θα ήταν το σωστό για τις συζητήσεις μας. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Διότι η οικονομική σύγκληση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μετά έχουμε ε, και περιφερειακές πτυχές. Η Λιθουανία εξαρτάται από την Πολωνία, τη Γερμανία. Υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν άλλες ιδιαιτερότητες το γραφείο να έχει τις δικές του. Θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι οικονομικές περιφερειακές πτυχές. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να δούμε αυτή την ε, διάσταση, την περιφερειακή. Πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την οικονομική σύγκληση και σήμερα δεν αφιβάλλει κανείς ότι υπάρχει ένας διάλογος αλλά πρέπει να ενισχυθεί. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το πράξουμε και με ποιο κόστος. πού, πόσες φορές θα συναντηθούμε ετησίω. Ίσως να προσφύγουμε σε τηλεδιασκέψεις για να αποφύγουμε ε, τις πτήσεις που σημαίνουν και περαιτέρω κόστος. Τώρα, μόλις αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της, Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Ε, εμείς να πω ότι συζητήσαμε τη στρατηγική της Λισαβόνας. Συζητήσαμε πολύ καιρό. Αλλά αποτύχαμε. Τώρα αρχίζουμε την ε, πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να συζητήσουμε τεχνικές πτυχές γιατί ξέρουμε, ο διάβολος στη λεπτομέρεια κρύβεται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να επιμένουμε ο διάλογος μας θα πρέπει, αυτό επιθυμώ, να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένος. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στην Ιταλία και πάλι. Παρακαλώ, κύριο Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πολλές φορές αναφέρθηκε σε προηγούμενες ευκαιρίες και συναντήσεις και η Ιταλία ανέκαθεν ναι, συμμεριζόταν την πρόταση του κ. Λαμασούρ για ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους θεσμούς. Θα ήταν χρήσιμη μία συνάντηση ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ώστε να επαληθεύουμε πριν ή μετά από τους εθνικούς προπολογισμού αν ε, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έγινε σεβαστός και οι υποδείξεις του έγιναν σεβαστές στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να αφορά τη σύγκληση των οικονομικών πολιτικών για την υλοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020. Η πρόταση Λαμασούρ προβλέπει μια συνάντηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πριν από την έναρξη των της εξέτασης του προπολογισμού δηλαδή το Σεπτέμβριο για την Ιταλία. Να δούμε δηλαδή αν οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ανάπτυξη, παιδί κτλ. και όλα αυτές οι υποδείξεις έχουν γίνει σεβαστές στον εθνικό προπολογισμό. Θα πρέπει η εθνική κυβέρνηση να παρουσιάσει επισήμως τον προπολογισμό. Το σημείο κλειδί είναι το περιθώριο ελιγμού, όπως ανέφερε και προηγουμένως η συγγήτρια και συνάδελφος Ζουρζέτη, από τη, ο συνάδελφος από το Κοινοβούλιο. Για την περασμένη χρονιά έχουμε έλλειμμα 4,6 σε σχέση με το 5 που είχε αρχικά προβλεφθεί και η ανάπτυξη του ΑΕΠ ήταν 1,3 χωρίς όμως οποιαδήποτε παρέμβαση ή κίνητρο από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Ωστόσο σήμερα ο προπολογισμό με μετρά κατά το 1,20 αυτή τη στιγμή. Ίσως να αυξηθεί το στο μέλλον, αλλά για την ώρα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή το να δοθούν περισσότεροι πόροι για την έρευνα σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν ε, πόροι, για παράδειγμα, από την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι η έδρα διακοινοβουλευτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελεί την ευκαιρία για να επαληθεύσουμε το βαθμό σύγκληση κάθε χώρα προ κοινού ευρωπαϊκού στόχου, για να αποδειχτούν και οι ενδεχόμενες δυσκολίες της χώρας στη διαδικασία σύγκλησης αλλά και επίσης για να διευκολύνουμε με μονομένα εθνικά κοινοβούλια να προβούν σε επιλογές που αυτές τις περιόδους είναι εξαιρετικά δύσκολες και οδυνηρές. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Όλα Σμιτ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you very much, Madam Chair. Uh, eating sandwiches is of course... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε για τα σάντουιτς και τα σάντουιτς τρώμε όλοι. Αλλά εγώ φοβάμαι σε λίγο θα έχουν τελειώσει και τα σάντουιτς. Θα μας τα έχουν φάει οι Κινέζοι και κάποιοι άλλοι. Και αυτή είναι ίσως μία από τις βασικότερες προκλήσεις σήμερα. Το λέω αυτό με κάθε ταπεινοφροσύνη, διότι πιστεύω ότι είναι μόνος τρόπος ε, η συνεργασία για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Βεβαίω είναι δύσκολο. Έχω διατελέσει μέλος και της Σουηδικής Βουλής και τα γνωρίζω αυτά. Ξέρω πού είναι τα όρια και οι γραμμές ε, των κυρίαρχων κρατών. Αλλά κάθε μέρα μετακινούνται αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε αυτό που σήμερα συμβαίνει στην Ιαπωνία μας επηρεάζει όλους. Μπορεί να μην το θέλουμε, να μην το επιθυμούμε, αλλά συμβαίνει αυτό. Και οι Lehman ε, Brothers και κάποια κακά δάνεια που δώσανε στο Κάνσας μας επηρεάζουν βεβαίως. Και είναι απορία άξιο γιατί έχουμε σήμερα τόσο πρόβλημα να δούμε μέχρι πού μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει όριο στη συνεργασία κυρία Βίκη Φόρτ. Μέχρι το άπειρο. Ακόμα και στο Λονδίνο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας τα προβλήματά σας. Θα μας δοκιμάσει η ιστορία και θα έρθουν να μας ζητήσουν και τα ρέστα. Αυτό δεν είναι νομοθεσία περί διαζυγίων. Δεν είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. δεν είναι ένα θέμα ίσονο σημασία νομικό, είναι πώ θα διατηρήσουμε τα κράτη μα. Αλλιώ θα χαθούμε. Η Παρασκευή είπαν για το σύμφωνο αυτό ότι στις 24 και 25 Μαρτίου θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μας πούν τα κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη αν θέλουν να συμμετέχουν στο σύμφωνο. Ναι ή όχι, είσαι μέσα ή είσαι έξω. Τόσο απλό. Και κατά τη δική μου άποψη που προέρχομαι από μια χώρα εκτός του ευρώ και πραγματικά θέλω να μπω στο ευρώ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα διχάσει την Ευρώπη. Θα τη διχοτομήσει για να μην πω ότι θα την τριχοτομήσει. Και είναι δική μας ευθύνη να πούμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε, μπορεί να είναι αυτό και σταδιακά, αλλά βασικό μα στόχο είναι να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία θα συνεργάζεται με έναν τρόπο στιβαρό και ε, βιώσιμο. Ευχαριστώ. Και τώρα από τη Λετωνία, ο κύριος Ρίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ κι εγώ ε, σε αυτά τα θέματα και να συμμετέχω στην τόσο ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Να σας πω τι γίνεται στη Λετωνία για το προπολογισμό μας και να σας δώσω και μια ιδέα για το μέλλον. Μέχρι τώρα έχουμε το πρόγραμμα ε, σύγκλησης που δεν συνδεόταν πάρα πολύ με τον προϋπολογισμό. Έχουμε ένα ετήσιο προϋπολογισμό και ένα πολιετές ε, σχέδιο, ένα πολιετή σχεδιασμό, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέχρι στιγμής ε, ευρωπαϊκές. Γι' αυτό είναι και πιο βαθιά η κρίση όμως, διότι δεν έχουμε αυτή τη σύνδεση. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει σε μια ισορροπία αυτή την εθνική πτυχή με την ευρωπαϊκή. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι τα κράτη είναι πολύ στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και προβλήματα σε μια γειτονική χώρα μπορεί ε, να οδηγήσουν σοβαρή οικονομική κατάσταση ε, ανετική στη Λετωνία και το αντίστροφο. Εμείς υποστηρίζουμε πολύ την τη σύνδεση του εθνικού προπολογισμού με τον ευρωπαϊκό και την παρακολούθηση αυτού. Είναι λογικό. Τα εθνικά προγράμματα και τα προγράμματα σύγκλησης ε, καταρτίζονται από κοινού κανονικά. Έτσι λοιπόν, στη Λετωνία πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα σύγκλησης και ο εθνικός προϋπολογισμός είναι ε, δεκτά και τα δύο στο Κοινοβούλιο και εξετάστηκαν και σε επιμέρους επιτροπές, ε, διαρκείς επιτροπές της Βουλής μας. Η κατάρτιση του προπολογισμού έχει μείνει πίσω πρέπει να σας πω φέτος, γιατί ε, πρώτα υπήρξε ένας διορθωτικός προπολογισμός για το 2011, αφενός αυτό και αφετέρου θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημοσιονομική μας πειθαρχία και αυτό να κατοχυρώνεται και στους νόμους μας. Χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερο χρόνο. Το χρονικό πλαίσιο που μας ε, προτείνεται με αλφαγιώτα έχει διάφορα στάδια και για τα προγράμματα σύγκλησης και συνοχής. Δεν οκληρώνονται όλα ταυτόχρονα. Υπάρχει ένα περιθώριο ενός μηνός. Δεν ξέρω αν χρειάζονται ειδικέ ε, διαδικασίες για μας. Ε, θεωρούμε ότι η δημοσιονομική πολιτική και ε, η χρηματοπιστωτική και για τον προπολογισμό είναι κάτι που παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και θα πρέπει να επιμείνουμε για να έχουμε ένα βιώσιμο σχέδιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, με τα εθνικά κοινοβούλια βάσει των ισχυών των νομοθετημάτων. Δεν χρειάζονται νέε διαδικασίες λοιπόν κατά την άποψή μας και σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, είναι πάρα πολύ σημαντική η ανταλλαγή εμπειριών. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω εδώ με τους προέδρους των επιτροπών που μίλησαν προηγουμένως. Δεν φτάνει μία συνεδρίαση ούτε δύο το χρόνο. Χρειάζονται περισσότερες, πιο τακτικές κοινέ συνεδριάσεις εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις, αλλά να συμμετέχουμε και στη διαδικασία συντονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Από τη Σλοβενία, ο κύριος Τσέπιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χθεσινή ομιλητές και η σημερινή μας ε, και η σημερινή εισήγηση του Πρόεδρου Ρομπόη γέμισαν αισιοδοξία ότι στην Ένωση Ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε να βγούμε από αυτήν την οικονομική και αναπτυξιακή κρίση με τρόπο που να μας ε, κάνει ακόμη πιο δυνατούς και έτοιμους για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι μια πολυπολιτιστική ήπειρος και δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν συντονίσουμε τις στρατηγικές μας ανάμεσα σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Οι θυσίε των πολιτών μας είναι πολλές και διάφορες και γι' αυτό η συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων με τα ε, ευρωπαϊκό είναι πολύ σημαντική. σημαντικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας είναι η σημερινή συνεδρίαση και θα ήθελα να γίνουν και περισσότερες τέτοιου τύπου συνεδριάσεις. Η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε διάφορα επίπεδα και γι' αυτό και η επιτυχία μας θα πρέπει να μετράτε βασικά σε σχέση με τον αδύναμο κρίκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση έδειξε ότι η έλλειψη σταθερότητα σε ένα από τα κράτη-μέλη μπορεί να υποσκάψει ολόκληρο το νομισματικό σύστημα. Και δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα σε σχέση με την ανάπτυξη ανήκει η προβληματική χώρα. Εμείς στη Σλοβενία ήδη έχουμε συντάξει ένα εθνικό πρόγραμμα το οποίο φυσικά βασίζεται σε ορισμένα σημεία κλειδιά που θα ήθελα να σας αναφέρω. Καταρχήν μακροοικονομική εποπτεία που περιλαμβάνει μακροοικονομικές προβλέψεις, ε, εκτίμηση των μακροοικονομικών επιπέδων ανάπτυξης, ε, παγιωμένη οικονομία από το 2011 μέχρι το 2015, αλλά και μέχρι το 2020 σε δεύτερη φάση, αλλά και ορισμένα μέτρα για την ε, επίτευξη των προτεραιοτήτων μας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης η Σλοβονία είχε επίσης υπερβολικό έλλειμμα πάνω από το 3% και στόχος μας είναι να επανέλθουμε στο ποσοστό 3% που θεσπίζεται από τη συνθήκη του Μάστριχτ και να έχουμε ανάπτυξη από το 2015 και μετά βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το διαρθετικό έλλειμμα, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των υπηρεσιών και να ε, καταργήσουμε τα εμπόδια στον επιχειρηματικό τομέα, να αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι το 3% του ΑΕΠ, δηλαδή μια επί του 3 αύξηση σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ε, επιτυχία μας και φυσικά μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας αλλά και περισσότερο συντονισμός ε, όσον αφορά τις πολιτικές ε, μισθών και παραγωγικότητας και γι' αυτό και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται να προβούμε σε μεταρρύθμιση της, της ανώτατης παιδείας και Επίσης, οι υποδομές ε, στις μεταφορές είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την οικονομική μας ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ μας. Ενεργειακή πολιτική, κοινωνική ασφάλιση και δημόσια διοίκηση μεταρρυθμίσεις εκεί, όλα αυτά φυσικά μεταφράζονται στον εθνικό μας προπολογισμό και η συνεργασία μας με άλλους, τη συνεργασία μας με άλλους φορείς όπως ε, και η Ένωση φυσικά. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Περβάνς Μπερές κάνει μια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Περβάνς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην αρχή, στην πρώτη μου παρέμβαση, ήμουνα κάπως συγκρατημένη. Αυτές οι ανταλλαγές απόψεως, απόψεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε εδώ και χρόνια. Η ιδέα ήταν να συζητήσουμε τις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής. Και το ανέφερα αυτό στην παρέμβασή μου στο, στην ε, συζήτηση με τον πρόεδρο. Ξέρετε, αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσει κανείς να κάνει μια διαγνώση και με βάση την οποία οι χώρες μέλη θα τακτοποιούν τα του προπολογισμού τους. Μου συνέβη στο παρελθόν να δω ποια ήταν η συζήτηση όσον αφορά τα του προπολογισμού σε κάθε κράτος μέλος. Έχουμε μια ε, αυτό που έχει να κάνει με κατευθυντήρια σε ευρωπαϊκέ γραμμέ, διαπιστώνω ότι ήταν κάτι το οποίο το κάνανε μόνο οι αντιπολιτευόμενοι σε κάθε χώρα. Δηλαδή, να μπορούμε, πρέπει να έχουμε μια από κοινού ε, συζήτηση πριν, νωρίτερα, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη διαφοροποίησεις από χώρα σε χώρα. Και, και είχαμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία μας οδήγησε σε ένα διέξοδο και φτάνοντας στην ε, κατάσταση του ευρώ έχουμε μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε αποκλήσεις. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό ε, νόμισμα και αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε συγκλήσεις. Σήμερα ξανά βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το θέμα με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτό που θέλουμε είναι να μην ξαναγίνει το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι από μια χώρα η οποία ήταν τη πρώτη που είπε να έχουμε μια οικονομική διακυβέρνηση. Απ' τη μια λένε αυτό και απ' την άλλη όμως ε, την άλλη όμως έβλεπες και στη χώρα μου ότι οι Βρυξέλλες δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν. θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι, ανοιχτοί, να από κοινού να κάνουμε μια διάγνωση, να λάβουμε υπόψη τις διαφοροποιήσει και να καταλήξουμε στο τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Από κοινού θα πρέπει να συζητήσουμε, να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ συμμετέχω σε αυτή τη δικασία εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε μια πραγματική συζήτηση ανάμεσά μας. εγώ θα ήθελα να έρχεστε εσείς εδώ πέρα με τις δικές σας προτάσεις. Παρεμβάσεις να κάνετε. Να μην μακρηγορήσω φυσικά, αλλά θα πρέπει να δούμε την ουσία του πράγματος. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τώρα. Η Επιτροπή τον Ιανουάριο έχει κάνει ένα, ένα, ε, καταθέτει ένα έγγραφο το οποίο έχει να κάνει με την ετήσια οικονομική ανάπτυξη. Από αυτό το σημείο και μετά, αυτό εγκρίνεται το Μάρτι από το Συμβούλιο και πριν από το Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου, η Επιτροπή αρχίζει συζητήσεις με κάθε χώρα μέλος να δει ποιε είναι οι συστάσει στο σύνολο το, του προσανατολισμού αυτού όσον αφορά τη θέση κάποιας, κάθε χώρας. Ε, και θα πρέπει να κάνει τον δικό της χάρτη κάθε χώρα. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Είδα. Είδα. Ε, είδα την πρόταση που έκανε ο Γάλλος πρόεδρος του, της Ανασυνέλευσης. Ε, η πρότασή του οδηγεί, είναι, οδηγεί σε καθυστερήσεις. Θα πρέπει να έχουμε, να γίνει σαφές ότι πρέπει να έχουμε αυτό τον διάλογο προσανατολισμού. Στα πλαίσια του Κοζάκ, για παράδειγμα, υπήρξε μια εβδομάδα ευρωπαϊκή, κάτι το οποίο δεν πέρασε πολύ καλά, αλλά την άλλη θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αν θέλουμε όντως να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, να έχουμε πραγματικά μια συζήτηση για ποια είναι η οικονομική η ευρωπαϊκή πολιτική, χρειάζεται κάτι παραπάνω από δυόμιση μέρες. Θα πρέπει να δουλέψουμε, να δούμε κάποιο να αναλάβει τα θέματα που να κάνει με τον ιδιωτικό χώρο, κάποιο κάποιο άλλο θέμα. Και αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να περάσω. Χαίρομαι όμω, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό, διότι είμαστε σε μια καμπή θα έλεγα. Είμαστε σε μια εμβριακή κατάσταση. Πλέον γίνεται σοβαρό το θέμα του Ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει φυσικά να δώσουμε μια έμφαση ε, στην ευρωπαϊκή ζώνη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι πραγματικά αν έχουν και άλλες ιδέες κάποιοι συνάδελφοι μπορούν να μας τις διαβιβάσουν για τις εκθέσεις σου. Έχω άλλους δύο ακόμα από το Εθνικά Κοινοβούλια και μισή ώρα και ίσως θα θέλει να απαντήσει και το πάνελ. Λοιπόν, από τη Γαλλική Γερουσία, κύριος Πάτρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά. Θα μιλήσω στο ίδιο θέμα σε σχέση με αυτά που είπε η προλαλήσασα Ε, για τη διαδικασία αυτή, όχι τη η οποία ήταν πάρα πολύ σωστή. Η συνθήκη της Λισαβόνα έδωσε αρμοδιότητε στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, τότε σκεφτόμασταν περισσότερο την μικροκουρικότητα. Να ξέρει καθένα ποιε είναι οι αρμοδιότητε του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά σε εθνικό. Και η κρίση οδήγησε μια κατάσταση όπου τα εθνικά κοινοβούλια ψηφίσανε ούτως ώστε να ε, υπάρχουν κάποιες εγγύησεις όσον αφορά για, τις, για, τα, για το χρέος. Η Ευρώπη όπως είναι σήμερα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Οι αποφάσεις λοιπόν έπρεπε, ήταν θέμα αρμοδιοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων. Η, κρίση στο Eurogroup οδήγησε σε μια, ε, σε μια κατάσταση όπου έχουμε από τη μια τις, τα, τις που έχει να κάνει με, τα, με τους προπολιούς σε εθνικό επίπεδο. Φυσικά και έχουμε να κάνουμε με αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά όπως και να έχει κατάσταση θα ήθελα να πω ότι αυτό μας υπενθυμίζει ότι το καλύτερο θα ήταν να, να δουλέψουμε από κοινού. Εγώ είμαι από τη γερουσία της Γαλλίας και ξέρω ότι αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο και δύσκολο. Θα πρέπει να ξαναδούμε, να ξαναδούμε τη διαδικασία που έχει να κάνει με τον προπολογισμό. Η Σιλβί Μπουλάρ πριν από λίγο ανέφερε για τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν να κάνουν με τη διεύρυνση της συναπόφασης. Να δούμε δηλαδή πώς, θα έχουν, πώς έχουν τα πράγματα σε γενοτικό επίπεδο σήμερα και πώς ακριβώς θα ισχύουν στο μέλλον. Έχουμε υποχρέωση να μάθουμε να, να συνεργαζόμαστε από κοινού και ο καθένας μας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, θα πρέπει να ακούει να ακούει τους μεν και τους δε, να καταλαβαίνει τις ιδιαιτερότητες του καθένα, αλλά, αλλά, αλλά όπως, είναι, όπως ελέγχθηκε πριν, ο καθένας να, να μην δείξει ούτε υπεροψία, κατανόηση μάλλον και συνεργασία. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς σε ό,τι κάνουμε. Ο διάλογος είναι απαραίτητος και δεν θα είναι πάντοτε εύκολος. Επίσης θα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε από κοινού να το κάνουμε σοβαρά και επίσημα. Αλλά όπως η Περβάνς Μπερές πριν από λίγο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διάλογο καθημερινό. Να μάθουμε να δουλεύουμε από κοινού και συνέχεια. Δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται φαντασία και πραγματικά πολιτική βούληση. Αλλά θα είναι σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και μακροπρόθεσμα θα είναι σίγουρα καλύτερα έτσι για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και τώρα από το Βέλγιο η κυρία Γκέρκενς. Euh, Είμαι ευτυχής που παρεμβαίνω τώρα σε αυτή τη συζήτηση, διότι πιστεύω πως όλοι στο πλαίσιο του Βελγικού Κοινοβουλίου επιθυμούν να υπάρξει ένα πραγματικό σχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει μια κοινοτική μέθοδος εργασίας πέρα από την κυβερνητική μέθοδο. Αλλά είναι αλήθεια που και ο συνάδελφος Βαντιμπρούκ ε, το τόνισε πριν από λίγο ότι είναι σημαντικό για μας το πρότυπο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιτρέψει μια ισορροπία ανάμεσα στη, σε κοινωνικές, στην κοινωνική και την οικονομική διάσταση. Και Βρισκόμαστε σε μια καμπή με αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο με τις έξι συστάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση, ταυτόχρονα τη συζήτηση για τον πολιετή προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε μια φάση που θα χρειαστεί από κοινού το Κοινοβούλιο Εθνικό και Ευρωπαϊκά, ε, ευρωπαϊκ, συγγνώμη, Εθνικά και Ευρωπαϊκό να συνεργαστούμε και να δούμε πώς θα μετρήσουμε και πώς θα προσανατολίσουμε τις πολιτικές μας. Έχω την εντύπωση ότι για την ώρα μέσα σε αυτούς τους δείκτες που υποτίθεται ότι είναι της ανταγωνιστικότητας, διάφοροι δείκτες που αφορούν δαπάνες προς αποφυγή, πολύ λιγότεροι για τις ε, δυνατότητες εσόδων που θα μπορούσαν να έχουν τα κράτη και η Ένωση και λιγότερο ενδιαφέρον για το ποιον τρόπο θα βρούμε για να εξετάσουμε επενδύσεις σε υπηρεσίες ε, στην ε, υγεία, στην παιδεία, που θεωρούνται τομείς οικονομίας και πλούτου επίσης. Και εδώ νομίζω είναι σημαντικό να γίνει μια συζήτηση πριν και το πριν είναι τώρα στην ουσία και στις επόμενες εβδομάδες, γιατί θα πρέπει να γίνει συζήτηση πριν τα κράτη να υποβάλουν τα προγράμματά τους, που θα εξεταστούν επί τη βάση των δικτών που θα έχουν αποφασιστεί. και που θα μπορούσαν να είναι πολύ περιοριστικοί σε σχέση με την ισορροπία που αναζητάμε. Και για να απαντήσω στην Γαλλίδα ε, Ευρωβουλευτή που μίλησε πριν από λίγο ότι ανάμεσα στην πραγματική, τα στιγμές μάλλον πραγματική συζήτηση ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια είναι πολύ σημαντικά, σημαντικές συναντήσεις. Εντάξει, η ανταλλαγή γραπτών και επαφές ε, ε, εξ αποστάσεων, όμως αυτό δεν αντικαθιστά τη δυναμική της ε, πραγματικής επαφής ε, ώστε να υπάρξει κάτι το ζωντανό και πραγματικά να υπάρχει αλληλεπίδραση. Τουλάχιστον αυτό είναι το αίτημα το οποίο διατυπώθηκε εδώ και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να επαναληφθεί και στα εθνικά κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιους έξτρα ομιλητές. Να στραφώ στον Ιστβαν Τζόσα και μετά έχω και άλλον έναν ομιλητή από τη Γερμανία. Και μετά την Βίκη ε, Φόρντ. Αν θέλει κάποιο ακόμα, τώρα να ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Σάρων. Που μου δίνει το λόγο ε, ω συμπρόεδρο. Τα σενάρια εργασίας υπαγορεύονται από τη ζωή την ίδια. Η Ουγγαρία έχει ως πρόγραμμα για την Προεδρία ε, την ισχυρή Ευρώπη. Έρχεται όμως η ζωή και μας επιβάλλει ένα πρόγραμμα πολύ πιο ισχυρό. Αυτό το έδειξε και η συζήτηση. Είναι πραγματικά πολύ εύγλωτο το παράδειγμα. Στις 11 Μαρτίου λήφθη μια απόφαση πάρα πάρα πολύ σημαντική. Είναι με ε, απόφαση των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά τίθεται ένα ε, ουσιαστικό ζήτημα εδώ σε αυτές τις καλές αποφάσεις μπορούν να συμπεριληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης, τα υπόλοιπα, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης και τα υπόλοιπα 10 για να επωφεληθούν. Το είπε και ο κύριος Φανρόμποϊ στην αρχή. Το σύμφωνο για το ευρώ δεν είναι για να έχουμε ένα σύμφωνο, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά για να διαφυλάξουμε τα επιτεύγματα του κοινωνικού κράτους, όπως είπε και η προλαλή σας από το Βέλγιο. Να διατηρήσουμε το κοινωνικό και οικονομικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Είναι σημαντικό με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούμε προς ε, μια ισορροπία μεταξύ του οικονομικού σκέλους και του κοινωνικού. Σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Φόρτ, εγώ είμαι μαθηματικό στο επάγγελμα και εργάζομαι στον τομέα των θετικών επιστημών. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε η κυρία Φόρτ. Η οικονομική κρίση επιδεινώθηκε και εκεί διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο ε, το έργο κάποιων ταχυδακτηλουργών, γιατί δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Γιατί έτσι έδρασαν, σαν ταχυδακτηλουργοί. Και αυτό που χρειάζεται είναι πολύ σαφείς κανόνες, όχι τρίκ, τεχνάσματα και ταχυδακτηλουργίες. Και πολύ ε, σωστές διαδικασίες. Σαφείς, εμείς οι πολιτικοί μπορεί να έχουμε όλους τους ευγενείς στόχους που θέλουμε και τα μεγάλα ιδανικά, αλλά πίσω από την πλάτη μας διάφοροι μάγοι, ταχυδακτηλουργοί, ε, μαγειρεύουν σκοτεινά πράγματα. Άλλο σημαντικό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ότι χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των Πρωθυπουργών και Αρχηγών Κρατών ε, με βάση το σύμφωνο της 11ης Μαρτίου και σιγά σιγά να προσεγγίζει αυτό τις εθνικές ε, επιδιώξεις και τα εθνικά σχέδια. Αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Έχουν ιδιαιτερότητες οι χώρες, προφανώς. Αλλά είπαν πολλοί συναδελφοί ότι χρειάζεται κάποιο είδου σύγκληση. Δηλαδή, αυτό που εδώ και χρόνια κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την επικεφαλίδα πολιτική συνοχής είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε και όχι να το εγκαταλείψουμε, να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη συνοχή και τη σύγκληση. Και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία τώρα να προχωρήσουμε με ειλικρινή διάλογο. Και σαν να μην είχαμε αρκετή δουλειά στι πρωτεύουσές μα στα εθνικά κοινοβούλια χρειάζονται, όντως χρειάζονται περισσότερε συνεδριάσει και θα πρέπει να έχουμε πιο πολλή δουλειά και στη συνεργασία μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι κυβερνήσει καταρτίζουν προγράμματα δράση εθνικά και σχέδια, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα συνεννοούνται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την εκπροσωπούν από κοινοβουλευτική πλευρά μόνο οι ευρωβουλευτέ. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μα αυτό. Είναι και οι εθνικοί βουλευτέ. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ και τελειώνω ε, για τη σημερινή συνεδρίαση και ελπίζω να μην περάσει απλώς στην ιστορία η 11η Μαρτίου ως ημέρα ε, του συμφώνου για την Ευρωζώνη, αλλά να είναι και η αρχή μιας συνεργασίας ε, η σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Έρχονται και προστίθεται συνέχεια κάρτες. Νομίζω κάποια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρώνουμε. Βίκη, προτείνω να μιλήσει τελευταία γιατί έχει αναλάβει το πλαίσιο αυτό δεν μπορείς να συνοψίσεις. Ε, χάρηκα από αυτό που άκουσα για τα μαθηματικά. Έχουμε εδώ διάφορους τέτοιους ε, στην αίθουσα και συναδέλφους. Ο κύριο Μπίντινγκ τώρα από τη Γερμανία. Τώρα δεν ξέρω αν είχαμε συνεννοηθεί και εγώ μαθηματικός είμαι, αλλά και ηλεκτρολόγος. Και επειδή ε, ε ως τεχνίτης ε, μπορώ να χειρίζομαι κάποια πράγματα πολύ πρακτικά, ε, συνεχίζω από τον προαλήσαντα. Είναι πολύ σημαντική η σύγκληση, κοινωνική Ευρώπη, ισχυρή Ευρώπη, κοινωνική οικονομία τη αγορά. Διαπιστώνω όμω. και παρατηρώ ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αυξάνεται όλο και περισσότερο η φτώχεια ε, των κρατών ανά τον κόσμο με ε, συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια ιδιωτών και καταλήγουμε σε τέτοιες κρίσεις τεράστιες. Και τότε απαιτούν πάλι όλοι και περιμένουν από τα κράτη να ενισχύσουν τους ιδιώτες παρόλο που για την κρίση φταίνε σε πολύ μεγάλο βαθμό ιδιώτε. Από αυτά τα προϊόντα τα οποία τοξικά ονομάστηκαν και στη Γερμανία, ε, τα τοξικά παράγωγα, τα τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα. Προσοχή λοιπόν, να μην φτιάξουμε ένα σύστημα που να ενισχύει τη φτώχεια του κράτου και ταυτόχρονα τον πλούτο στα χέρια κάποιων ιδιωτών. Αν μιλάμε πρώτα για τι καταθέσει και τι αποταμιεύσει, είναι μόνο η μισή αλήθεια. Θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε ε, Μάλλον ε, για τον προπολογισμό λέμε να μειωθούν οι δαπάνε. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ενισχυθεί και ο τομέα των εσόδων. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσορίστηκε η ιδέα του τέλου στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτη και πριν από 10 χρόνια ε, δημιουργήθηκε η ΑΤΑΚ. Αλλά ε, ε κάποιος ε, επιμελής ε, χρηματιστής έκανε 50 ή 100 συμβάσεις την ημέρα αν δούλευε πολύ. Σήμερα κάνει 20 εκατομμύρια ε, συναλλαγές την ημέρα. Εκεί αυτό δεν πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Και τι γίνεται με τον πλούτο, με τη φτώχεια, πώς αποκλίνουν αυτά, πώς κατανέμεται, πώς αναδιανέμεται ο πλούτος. Γι' αυτό σκεφτόμαστε να βάλουμε και ένα φόρο ε, μεγάλης περιουσίας στη Γερμανία σε συνδυασμό με ένα φόρο κληρονομίας για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να φορολογεί το πλούτος και να δούμε τώρα εγώ περιορίζομαι στις χώρες της Ευρωζώνης να δούμε με ποιο τρόπο αυτοί που έχουμε ένα κοινό νόμισμα με τόσο διαφορετικές οικονομικές πολιτικές, κοινωνικές πολιτικές, δημοσιονομικές πολιτικές αν δεν καταφέρουμε μια καλύτερη σύγκληση τότε αυτό έρχεται σε αντίφαση με το ένα νόμισμα που έχουμε οι 17 όσοι έρθουν και, να συγκλίνουμε στο νόμισμα και να αποκλίνουμε στις άλλες πολιτικές. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα οδηγήσει σε κανένα καλό αποτέλεσμα και χρειάζεται νέα προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Now to... Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεπρού από το Βέλγιο. Δεκρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση που είχα, μικρή καθυστέρηση και ίσως αυτό που θα πω τώρα έχει καλυφθεί από προλαλήσαντες. Εγώ είμαι πολύ παλιό μέλος του Κοινοβουλίου. Ο καλός συνάδελφος Βαντεμπρούκ γνωρίζει ότι είμαι εκλεγμένος στη Βουλή 43 χρόνια, στη Βελγική Βουλή, 43 χρόνια. Παρακολουθώ όλη τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης εξευρωπαϊσμού διαφόρων πολιτικών, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που συμβαίνει όμως το τελευταίο διάστημα είναι ότι μιλάμε πάρα πολύ για το timing, για το χρονοδιάγραμμα, αλλά ξεχνάμε μία διάσταση που είναι πραγματικότητα σε πολλά κράτη-μέλη. Ξέρω ότι δεν μπορεί να σταθεί ένα κοινό νόμισμα αν δεν δούμε και την κοινωνική και την οικονομική ε, υποκείμενη βάση. Οι χώρες όμως διαφέρουν στην Ευρώπη μεταξύ τους. Ήδη από τον Ιανουάριο άκουσα για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής και τώρα είμαστε στο Συμβούλιο, στο Μάρτιο κτλ. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα ένα κορσέ για να συμμαζέψουμε λίγο τα δημοσιονομικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά. Συνεχίζω στα γαλλικά τώρα. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο ακόμα που θα πρέπει να προσθεθεί στη συζήτηση. Οι χώρες μας έχουν και εσωτερικές δομές ορισμένες, πάρα πολύ θεμητές και πάρα πολύ ιδιαίτερες, που σημαίνει ότι η εξουσία ασκείται σε διάφορα επίπεδα, είτε παράλληλα είτε ε, κάθετα. Είτε αυτή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Αυστρία είναι χώρες που έχουν δομές ομοσπονδιακές, με κοινότητες, με περιφέρειες, με οπόσποδα κρατήρια ή και με μεγάλες πόλεις που έχουν ε, μεγάλη σημασία από πλευράς προπολογισμού. Δηλαδή έχουμε ενότητες, έχουμε οντότητες διαφορετικές και πολλές φορές δεν ε, έχουν και συντονισμό μεταξύ τους γιατί είναι παράλληλες, έχουν ξεχωριστή οικονομική πολιτική, ξεχωριστή δημοσιονομική πολιτική δεν υπόκεινται σε καμία ανώτερη εθνική αρχή. Και οι χώρες αυτές, επαναλαμβάνω, θεμητά έχουν καταλήξει αυτά τα συστήματα. Τι θα γίνει, ε, πώς συγκεκριμενοποιείται αυτό το στοιχείο και οι συνέπειες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το θέτω αυτό προς συζήτηση στην καλή ε, αυτή αντιαλλαγή απόψεων. Ότι μπορεί να υπάρχει ένα στοιχείο χρόνου, ένα στοιχείο άρμοδιοτήτων και εξουσιών, ένα στοιχείο ιεραρχίας για τα έσοδα, για τις δαπάνες ή για το συνδυασμό και των δύο, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτό το στοιχείο της διάρθρωσης της κρατικής των διαφόρων χωρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος από το εθνικό Κοινοβούλια, ο συνάδελφος Μαρτίνς από την Πορτογαλία. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Είναι φυσικό και νομίζω όλοι συμφωνούμε γι' αυτό ότι χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό των πολιτικών και το ευρωπαϊκό εξάμενο ακριβώς αυτό είναι. Αλλά επίση συνειδητοποιούμε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα για την ε, ανταγωνιστικότητα απέναντι στην Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ. Σήμερα το πρωί, στο πρώτο είχαμε την εντύπωση ότι όσα είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι το εξή, ότι οι χώρες θα πρέπει να έχουν χρόνο για να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές. Όμως, ακριβώς αυτά τα σχέδια που οι ίδιες χώρες με την δική τους ευθύνη εφαρμόζουν είναι σκληρά μέτρα, μέτρα λιτότητας, όμως θα πρέπει να συνδυαστούν με το θέμα της προοπτικής ανάπτυξης, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα είναι όλο και πιο δύσκολα. Και οι χώρες δεν μπορούν να αφαιθούν μόνες τους, γιατί οι κερδοσκοπικές επιθέσεις ε, ε, είναι πολύ άριθμες και έντονες. Το θέμα λοιπόν της Ευρώπης είναι περισσότερη Ευρώπη μέσω αυτών των εργαλείων που εδώ εξετάζουμε Η Πορτογαλία δεν είδε την φούς και δεν είχε προβλήματα άλλα. Όμως είχε προβλήματα την ανάπτυξη, γιατί ήθελε να στηρίξει την καινοτομία, τις ε, δεξιότητες, διάφορες επενδύσεις για να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη ανάπτυξη της οικονομίας της και σε παραδοσιακούς τομείς όπως ε, στην υφαντουργία και την υποδηματοπία. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες δράσεις και η συζήτηση που είχαμε χθε το βράδυ με τον κύριο Τελόρ ήταν ε, παρόμοια, ότι μπορούσαμε να μιλήσουμε για την εφαρμογή ενός ε, φορολογικού μηχανισμού που να είναι ισότιμος και θα διευκόλυνε όλα τα κράτη-μέλη να ανατρέξουν στον ίδιο μηχανισμό. Θα ήταν κάτι στο οποίο θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Και να πω ότι η Πορτογαλία κάνει τη δουλειά της, ενισχύει και εναρμονίζει τους κανόνες ε, τους δημοσιονομικούς. Αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας, στην Επιτροπή Προπολογισμού και Οικονομίας, κάνουμε μια προσαρμογή ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τη σημασία της στήριξης ε, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε προϊόντα με μεγαλύτερη ε, προσθεθέμενη αξία. Αυτή την πορεία ακολουθεί η Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια και αυτό και αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία που υπάρχουν για την καινοτομία αλλά και για την δομή των πορτογαλικών εξαγωγών. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα επανέρχομαι στο Ευρωκοινοβούλιο και την Βίκη. Τι ωραίο να βλέπεις τόσους συναδέλφους μαθηματικούς εδώ. Καμιά φορά εγώ το πάω καλύτερα με τους αριθμούς παρά με τα λόγια. Ίσως γι' αυτό να παρανοούμε καμιά φορά. Με παρεξηγείτε. Βεβαίως κάθε χώρα μοιράζεται τις καλές πρακτικές της, και είναι ευπρόσδεκτα όσο γίνεται τα σχόλια για να μας βοηθήσουν όλους να ε, ε, δυναμώσουμε την προσέγγιση μας. Ούτε πρέπει να είναι ενιαία η προσέγγιση και η λύση, αλλά είναι συμπληρωματική. Το ξέρω ότι οι χώρες έχουν διαφορετικές ε, πραγματικότητες και διαφορετικές ε, μεθόδους και τραπούς μπορούν να ακολουθήσουν για να ε, ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Και επίσης αναγνωρίζω ότι υπάρχουν και χώρες στην Ευρωζώνη που μπορεί να θέλουν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο επίπεδο, πώς να το πω, συντονισμού, μη τι άλλο. Γι' αυτό περιμένω και τις προτάσεις για τα τεχνάσματα, τα χρηματοπιστωτικά των τραπεζών και τις ταχυδακτηλουργίες. Κανένας δεν θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτής της φούσκας στην Ιρλανδία ήταν τέχνασμα ή ταχυδακτηλουργία. Ούτε αυτά που λέει η ας πούμε, για τις πανικές τράπεζες που τις υποβαθμίζουν ε, πριν από λίγες εβδομάδες. Ούτε αυτό είναι ταχυδακτηλουργία. Είναι απλώς υπερδανισμός που έχει ε, ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ασίδωτος. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και μπορεί να υπήρξαν μαγειρέματα σε κάποιους εθνικούς προϋπολογισμούς για τις τράπεζες, για τη δυνατότητα, για τη ρευστότητα και την ευρωστία των τραπεζών. Βεβαίως χρειάζεται έλεγχος και στις ε, τράπεζες και για τη Βασιλεία, τα λέει η έκθεσή μου. Ένα παράδειγμα να δανειστώ μόνο. Στη δική μου έκθεση Ζήτησα από τα κράτη-μέλη, αν γίνεται, να μου υποβάλουν αυτό το θέμα. Ε, έχουν ανεξάρτητους ε, οργανισμούς που κάνουν προβλέψεις για τα δημοσιοοικονομικά. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και ότι χώρες το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα από εσά. Εγώ προτείνω να υπάρχει κάποια στοιχειώδης, ανεξάρτητη εποπτεία για να αποφύγουμε αυτά τα τρίκ και τα χειδακτηλουργίες και ζητώ στην Ευρωζώνη να είναι αυτό υποχρεωτικό και δεσμευτικό. Ε, αλλά νομίζω ότι συνιστάται και για όλες τις χώρες. Ε, για να βρούμε τη σωστή διατύπωση σας παρακαλώ κάντε προτάσεις για μια ανεξάρτητη εποπτεία ε, αυτών των θεμάτων. Με χαρά ε, να ακούσω ό,τι έχετε να πείτε μετά τη συνεδρίαση αυτή από τις διάφορες χώρες σας. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανένας άλλος το λόγο από το πάνελ, καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη συζήτηση σήμερα το πρωί. Θα μπορούσα να κάνω μερικά καταληκτικά σχόλια τώρα. Πρώτον, συνεχίζοντας από αυτά που μόλις είπε η Βίκη. Στο δημοσιονομικό πλαίσιο θέλουμε να ρίξουμε φως σε κάποιες σκοτεινές γωνιές που υπάρχουν ακόμα. Και αυτό ισχύει και για τους εθνικούς λογαριασμούς. Στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό της δέσμης ε, μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση προσπαθούμε να συνενώσουμε τα διάφορα μέσα, τα διάφορα εργαλεία που έχουμε. Είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είναι οι ασωματωμένες κατευθυντήρες γραμμές και για την απασχόληση αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη και έχουμε και το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και τη δέσμη μέτρων. Νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε πάλι στα μαθηματικά και να πούμε ότι θα πρέπει κανείς να καταλαβαίνει ε, τα διάφορα ε, ολοκληρωμένα, ολοκληρώματα στα μαθηματικά για να τα ενσωματώσει όλα αυτά. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε και την ένταση και, τη, ε, και το ρυθμό ε, των επαφών που έχουμε και περισσότερε συνεδριάσει, αν θέλετε να κάνουμε και ομάδε εργασία και να επανερχόμαστε στη συνέχεια να συνοψίζουμε. Πάντως έχουμε καταλάβει ότι τώρα στην οικονομική διακυβέρνηση συμμετέχουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο πρωτοφανή που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν και καλό είναι να συντονιζόμαστε και να συνεργαζόμαστε για να ακούγονται στο κάτω-κάτω οι φωνές των πολιτών περισσότερο και να ακούν και εκείνοι περισσότερο τους βουλευτές τους είναι πολύ σημαντικά όντω αυτά τα θέματα και θα πρέπει να τα προωθήσουμε. Θα διακόψουμε τώρα και θα ε, συνεχίσουμε στην ίδια αίθουσα στις 3 και 4. Από τις 3 και 4 λοιπόν μέχρι τις 5.30 ε, ε, θα είναι η απογευματινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα λέμε το απόγευμα.